Good afternoon, Reverends. Um, Καλησπέρα, σεβασμότατοι κυρίες και κύριοι, αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ασύνηθες μεν μια συνεδρίαση να ξεκινά σχεδόν στην ώρα της, όμως θα ξεκινήσω σχεδόν στην ώρα μου. Είστε όλοι άκρως ευπρόσδεκτοι στη σημαντικότατη αυτή διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και χαίρομαι που μπορώ να σας καλωσορίσω όλους. Όπως ξέρετε είμαι υπεύθυνη για τα θέματα του άρθρου 17 Μεγάλη τιμή για μένα να είσαστε τόσοι πολλοί εδώ και να μπορείτε να συμβάλλετε στη συζήτηση που είναι σημαντική και αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Κάποιες λεπτομέρειες οργανωτικής φύσεως. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για τους συγκεκριμένου και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που θα παραστούν. Υπάρχουν τα έγγραφα στα αγγλικά και στα γαλλικά και αν χρειαστείτε βοήθεια σας παρέχεται. Υπάρχει διερμηνία στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, πολωνικά, ελληνικά, φιλανδικά και ουγγαρικά, ουγγρικά συγγνώμη. Επίσης μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο η εκδήλωση. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη όταν σας καλώ να λάβετε το λόγο. Και έχουμε και επίσημους φωτογράφους που καλύπτουν την εκδήλωση και καλύπτουν τη συζήτηση. Τιμή για μένα που σας κάλεσα εδώ και σε πρώτερες συζητήσεις με εκείνους που επίσημα είναι εδώ να κάνουν παρουσίαση, θέλω να πω ότι με ενέπνευσε ενθουσιασμός από την ατμόσφαιρα της συνάθρησής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι θέλετε να είσαστε εδώ και να συμβάλλετε και εμείς στο Κοινοβούλιο και ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς επίσης επιθυμούσαμε διακαώς να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Είναι καλή αυτή η αρχή και χαίρομαι που ο πρόεδρος κ. Σταγιάννη που μας στέλνει χαιρετισμού και είναι εδώ το πνεύμα τη, μου ζήτησε να αναλάβω εγώ τις εργασίες του άθου 17. Πρέπει να καλύψω τη θέση του είναι πολύ δύσκολο. Είχε αυτό το ρόλο. Εγώ μαθαίνω και εργάζομαι σκληρά του ώστε να είναι καλό ο διάλογό μα. Ευχαριστώ και πάλι, Αντιπρόεδρε, κύριε Τίμερμαν. Συνεργαστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε παρόμοιο διάλογο με διακοσμικέ ε, οργανώσει, φιλοσοφική συζήτηση. Και τώρα εδώ κάνουμε ευρύτερη συζήτηση στα πλαίσια του άρθρου 17 και εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούμε. Άριστα, χρειάζεται στενή συνεργασία αυτό το θέμα και χαίρομαι μπορώ να πω ότι αυτό συμβαίνει. Έχουμε διαφορετικούς ε, ρόλους, αλλά πιστεύω στο ότι ισχύει ενώση ισχύει. Και αυτό εδώ αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος η συνάντηση αυτή από όταν διορίστηκα, συνάντησα πολλού από εσά και πολλού ηγέτε θρησκευτικών κοινοτήτων. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη συνάθρηση όπου εσεί είσαστε στη θέση του οδηγού και εμεί θα σα ακούσουμε. Το θέμα είναι το μέλλον τη Ευρώπη και ξέρω ότι είναι κάτι που εμεί τα θεσμικά όργανα το συζητάμε, το επεξεργαζόμεθα και σίγουρα στι κοινότητέ σα και εσεί σκεφτόσαστε και προβληματιζόσαστε για το είδο τη Ευρώπη που θα θέλατε και τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στο Κοινοβούλιο να σας πω ότι θετήσαμε δύο ουσιαστικέ εκθέσεις και αυτό είναι η συνεισφορά μας στη συζήτηση. Οι συνάδελφοι Μπροκ, Μπρεσό και Βερχόφστατ ετοίμασαν τι εκθέσει και τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Λευκή Βίβλο για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Χαίρομαι ιδιαίτερω διότι ήταν εφικτό να προετοιμάσουμε το σημερινό σεμινάριο σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και καλωσορίζω και ευχαριστώ τον προ... την, Τανούτα Χούμπνερ, την κυρία Τανούτα Χούμπνερ, την πρώτη τη Επιτροπή αυτέ και του δύο συνεισηγητέ, την κυρία Μπρεσό και τον κύριο Μπροκ. Διότι και αυτή ήταν σημαντικό κομμάτι των συζητήσεών μα και τη συναντήσεώ μα. Όπω γνωρίζετε, υπάρχουν πολλέ εκκλήσει μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και προέρχονται και εκ των έσω και των έξω και χρειάζεται σοβαρή μεταρρύθμιση. Αν θέλουμε οι πολίτε μα να μιλάνε για την Ευρώπη με έναν τρόπο με τον οποίο κουβεντιάζουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί σε ηγετικού ρόλου. Δεν αρκεί να πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα οι ηγέτε. Θα επιβιώσει η Ευρώπη μόνο μέσω τη ενέργεια και του ενθουσιασμού των λαών. Των λαών που ζουν στην Ήπεθρο, στα χωριά, ε, στι πόλει, στι μεγάλε πόλει τη Ευρώπη. Να καταλάβει ο κόσμο περί τίνο πρόκειται. Τι εννοούμε όταν λέμε Ευρώπη. Και το άρθρο 17 που διέπει αυτόν τον διάλογο έχει πλαισιωθεί το τρόπο. Και ο λόγο για τον οποίο είμαστε τόσο ικανοποιημένοι που σα φιλοξενούμε και σα ακούμε είναι ε, διότι και εσείς ε, έχετε ηγετική θέση στις κοινότητές σας και δεν είναι μόνο μια διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους αυτή. Αυτή είναι κάποια ψυχρή διατύπωση, να το πούμε έτσι. Ε, το πνεύμα του κατά τη συνθήκης είναι τέτοιο. Δηλαδή συζητάμε την καρδιά και την ψυχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Αυτό θα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Οι δυτικοί πατέρες Θέλαν να δημιουργήσουν μια ένωση που βασίζεται στι αξίε. Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη τη. Και οι φιλοσοφικέ οργανώσει και θρησκείε θέτουν τα μεγάλα ερωτηματικά. Προσπαθούν να σχηματίσουν την ευρύτερη εικόνα. Θέλουν να εργαστούν για το κοινό καλό, εντοπίζοντα τι θεμελιώδει αξίε και αρχέ που στηρίζουν τι κοινότητε μα. Η Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο από την οικονομία. Ε, είναι κάτι παραπάνω από ποσοστά και στατιστικά στοιχεία. Οι διαβουλεύσει σχετικά με το ποια μορφή θα θέλαμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον αφορά περισσότερο ε, την κοινή άποψη για τον κόσμο. Μια διαδικασία που δεν μπορεί να είναι απλώς ένα εγχείρημα τεχνικής φύσεως ή απλοί υπολογισμοί και διοργανώσεις θεσμών και προπολογισμών. Αυτά είναι σημαντικά θέματα αλλά δεν δημιουργεί το άθροισμά του στο σύνος Ευρώπης. Ευρώπη. Στι του Κοινοβουλίου λέμε ότι πρέπει να είναι όλο και πιο στενή η ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Και αυτός ο σκόπος τη Και ελπίζουμε ότι οι θρησκευτικοί και φιλοσοφικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλλουν στη δημόσια συζήτηση υπογραμμίζοντα τα κοινά στοιχεία των λαών της Ευρώπης, ξεκινώντα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του καθενό ανθρώπου. Οι πολίτε πρέπει να είναι στο επίκεντρο του όλου και θα πρέπει συνεχώ να διερωτώμεθα κατά πόσο πραγματικά ακούμε ε, αυτά που μα λένε οι πολίτε για το είδο τη Ευρώπη που θα ήθελαν να έχουν και να ζουν εντό τη. Τι περιμένω από την Ευρώπη να κάνει, να τι βοηθήσει την καθημερινή του ζωή και να βοηθήσει του άλλου. Το Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει σχετικά με αυτό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότατα και άλλα εργαλεία και μέσα, ώστε να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτε στην συμμετοχική δημοκρατία. Οι Ευρωπαίοι πολίτε και η σχετική πρωτοβουλία των πολιτών τη Ευρώπη δεν ήταν τεράστια επιτυχία και εξετάζεται. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα για την πρωτοβουλία και πώ μπορεί να αλλάξει και πρέπει να δούμε πιο πέρα τι γίνεται, να δούμε μέχρι το 2025 πώς θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία στο μέλλον, μαζί με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Τίμερμανς και τους συναδέλφους και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Όπως σας είπα, ακούμε, είμαστε σε θέση ακοής. Θέλουμε να ακούσουμε αυτά που ε, θέλετε να μας πείτε και να συναθρήσουμε τις συνεισφορές που ελπίζουμε ότι θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη συζήτηση περί του μέλλοντος της Ευρώπης. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας, για την προσοχή σας και καλό τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Τίμερμανς να μας ε, μιλήσει. Είστε πρόσδεκτους. Ευχαριστώ πολύ Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε να παραστώ σε αυτή τη συνεδρίαση όπως είπα την περασμένη εβδομάδα. Ήδη είχαμε άκρος καρποφόρα συνάντηση ε, με, κοσμικής, με κοσμικές ε, οργανώσεις και ελπίζω να έχουμε και άλλη συνάντηση με θρησκευτικέ οργανώσεις αργότερα στο έτος, νομίζω αρχές Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου, και για μένα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν θεσμικό όργανο είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι συναντήσεις. Δυστυχώς ε, την τελευταία δεκαετία και λίγο περισσότερο στην Ευρώπη αρχίζαμε να συγχέουμε μέσα και εργαλεία και στόχους. Ε, καμιά φορά η εσωτερική αγορά παρουσιάζεται σαν ένα ε, αυτοσκοπός. Καμιά φορά το κοινό νόμισμα θεωρείται αυτοσκοπός. Αυτά όμως δεν είναι τίποτα άλλο από εργαλεία, από μέσα για τη στήριξη των αξιών μας, των κοινών, των Ευρωπαίων, σε ένα πλαίσιο μακράς, πολύ μακράς ιστορίας συγκρούσεων, αντιπαράθεση στην Ευρώπη. Να μην συνομιλούμε, αλλά να πολεμούμε ένα τον άλλον, να μην πετυχαίνουμε συμβιβασμού, αλλά να θέλουμε να κυριαρχούμε ένα τον άλλον. Και την περασμένη Παρασκευή ήμουνα στην Έση, ε, όπου είχαμε θεατρικό φεστιβάλ και υπήρχε ένα έργο για τον Μαρτίνο Λούθυρο, Εορτάζοντας τα 500 χρόνια της μεταρρύθμισης, ε, βλέποντας λοιπόν το έργο και ακούγοντας στα λεγόμενα, θυμήθηκα ότι μια απλή έκκληση για αλλαγή, για μεταρρύθμιση, αν δεν γίνει αντιληπτή σαν πραγματική τέτοια έκκληση για μεταρρύθμιση, μπορεί να θεωρηθεί σαν με τοπική επίθεση κατά της καθιστικίας τάξεως και των θεσμών. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλυσίδα αντιδράσεων ε, που δεν ήταν αυτό που επιδίωκε ο Λουθύρο, αλλά ούτως ή άλλως συνέβη. Και μετά το θάνατό του η Ευρώπη ε, επί 100, 102 χρόνια, για να είμαι ακριβή, πριν βρούμε ισορροπία μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων, είχαμε χρόνια αιματηρών συγκρούσεων, θρησκευτικών πολέμων που κατέστρεψαν πάρα πολλέ ζωέ. Αυτή είναι η κοινή μα ιστορία και τώρα Είμαστε καθισμένοι εδώ γύρω από ένα τραπέζι με ανθρώπου που στι συλλογικέ του μνήμε γνωρίζουν την ιστορία τη συγκρούσεω και τη αντιπαράθεση στην Ευρώπη. Είχαμε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ χριστιανών. Ακόμα χειρότερα, αιώνε επί αιώνων αντισημιτισμού. Ε, και ήταν από οι τράγοι οι Εβραίοι, όποτε κάτι πήγαινε στραβό στι κοινωνίε μα, οδηγούσε στο να φοβούνται κάποιοι άνθρωποι και να είναι αβέβαιοι για το μέλλον. Είχαμε το σχετικά νέο φαινόμενο ε, του μίσου κατά των μουσουλμάνων που αυξάνεται σε πολλά κράτη-μέλη. Το συμπέρασμά μου είναι το εξή. Όποτε ο φόβος είναι κυριαρχο, κυρίαρχος παράγων στην κοινωνία, είναι εύκολη η χαλινά αγώγηση. Ο φόβο οδηγεί στην οργή, η οργή οδηγεί στην προσπάθεια εξέβρεσης ε, αποδιοπομπαίων τράγων και αυτή είναι η θλιβερή κατάσταση που οδηγεί σε πολέμου τελικά. Αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα αφορά ε, κάτι περισσότερο από την κοινή αγορά και το ευρώ. Αφορά το να βοηθήσουμε του Ευρωπαίου να μην στρέψουν ποτέ στις παρελθούσες αυτές συγκρούσει και του πολέμου. Και καμιά φορά υποτιμούμε αυτή τη θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασία με όλα όσα κάνουμε λάθος και θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν και θα πρέπει να αλλάχθούν με όλες τις ε, βελτιώσεις ε, που απαιτεί το κοινό μας εγχείρημα. Βελτιώσεις που θα επέλθουν αν συμμετάσχετε πλήρως στους διαλόγους θα πρέπει να παραμένουμε σε επαφή με τις θεμελιώδεις αρχές, τη θεμελιώδη αρχή, ότι αυτό το εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα ειρήνης, πρωτίστως εγχείρημα ειρήνης και χρησιμοποιούνται εργαλεία για να επιφέρουν την ειρήνη και εκεί να λειτουργεί η κοινή αγορά και το κοινό νόμισμα. Το λέω αυτό και σε μια εποχή όπου βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη ότι αισθανόμαστε εξαιρετικά άνετοι τη συνοδεία ανθρώπων που είναι σαν και εμάς. Και επιδιώκουμε διάλογο με ανθρώπους με τους οποίους ήδη συμφωνούμε. Και χάσαμε την τέχνη του διαλόγου με εκείνους με τους οποίους διαφωνούμε. Και ο μόνος τρόπος σε μια επικοινόμορφη κοινωνία όπως είναι δική μας, που μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινή αντίληψη των κοινών αξιών, είναι να μην αποφύγουμε τη συζήτηση με εκείνους με τους οποίους δεν συμφωνούμε. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να πετύχει ένα συμβιβασμό είναι να ακούσει εκείνους με τους οποίους διαφωνεί, όχι μόνο να ακούει εκείνους με τους οποίους συμφωνεί. Και νομίζω ότι έχουμε μακρά εμπειρία τώρα, ε, κυρίως όσον αφορά τους σκεφτικούς φορείς, να βρίσκουμε τόπους συναντήσεως όπου εκεί υπάρχει περιθώριο διαφωνίας, χώρος διαφωνίας και κοινών έδαφος. Αυτή είναι η ουσία πιστεύω για το πώς διοργανώνεται η Ευρώπη και πώς λειτουργεί η Ευρώπη όταν είναι στα καλύτερά της. Και νομίζω ότι έχουμε συλλογική ευθύνη να μην αποφεύγουμε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Ακόμα και ε, έχουμε βαθιές διαφωνίες. Είναι πολύ εύκολα μιλάμε για τους λαϊκιστές, τους ριζοσπαστικούς κλπ. Αλλά μας ενδιαφέρει πραγματικά γιατί οι άνθρωποι ψηφίζουν αυτούς τους ριζοσπαστικούς πολιτικούς, γιατί ακολουθούν ανθρώπους με αυτές τις ιδέες Εάν τους μιλήσουμε ίσως ανακαλύψουμε γιατί και ίσως εκπλαγούμε αν μάθουμε τα πραγματικά αίτια και ίσως να βρούμε και κοινό έδαφος, κοινό τόπο. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι κάτι του σήμερα είναι ανέφικτο. Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος ουσιαστικά σαν απότερο σκοπό έχει την εξέβρεση κοινού εδάφους, κοινού τόπου, να ακούμε ένα τον άλλον. Ο Αλμπέρ Καμίσο έλεγε ότι το μόνο που διακρίζει εμάς από τα ζώα είναι η δυνατότητα να βλέπουμε μέσα από τα μάτια του άλλου. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ικανότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιώδης για να βρούμε διέξοδο από τα σημερινά προβλήματα. Όλοι είμαστε ηθικάοντα. Ε, κανείς δεν έχει το μονοπόλιο του σωστού. Ούτε έχει κάποιος το μονοπόλιο όσον αφορά το τι είναι εσφαλμένο. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι προσπαθούμε να είμαστε ηθικοί άνθρωποι όσο μπορούμε. Εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος γι' αυτό και μπορούμε όλοι αυτό να το επιτύχουμε αν αστερνιστούμε το διάλογο σαν έναν τρόπο προωθήσεως του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Γι' αυτό και το κοινό μα σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια λευκή βίβλο η οποία δεν είναι πλέον πατανιστικό τρόπο προσεγγίσεω των πραγμάτων και παρουσιάσεως ενός ε, σχεδίου πλήρου, για να πούν οι αποδέκτες ναι ή όχι αλλάξτε αυτό ή εκείνο παρουσιάζει διάφορες επιλογές, διάφορες κατευθύνσεις που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ευρώπη ε, τα επόμενα έτη, οι γενιές ακόμα, και είναι ένα έγγραφο ανοιχτό για διάλογο με τα κράτη-μέλη. Και εδώ των κρατών μελών ελπίζουμε οι κυβερνήσει να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία του ώστε να ξεκινήσουν διάλογο με του πολίτε όσον αφορά την κατεύθυνση κοινή Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτή είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό εκείνοι που, αντικα... που προβληματίζονται επί θεμάτων και τώρα να βρω ένα κοινό παρονομαστή μεταξύ φορέων θρησκευτικών και μη θρησκευτικών είναι προβληματισμό προβληματισμός περί του ανθρώπου και της θέσεως αυτού στην κοινωνία επί ηθική Εάν δεν προβληματιστούμε περί της Ευρωπαϊκής Ενώσεω ξεκινώντα από ηθικέ ρίζες δεν έχει νόημα γι' αυτό πιστεύω, αυτό το ρόλο θα παίξει ο διάλογός μας στα πλαίσια του άρθρου 17 και είναι σημαντικός για όλους μας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Ζητώ συγγνώμη πρέπει να αποχωρήσω νωρί. Πρέπει να πάω σε μια άλλη δημόσια εκδήλωση αργότερα στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ και θα αποχωρήσω το πρωί, θα φύγω το πρωί πολύ νωρί να πάω στην Ελβετία να συζητήσω το θέμα της Κύπρου αλλά για μια ακόμη φορά θα ήθελα να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε, να βρούμε κοινέ απαντήσεις για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι γενιές μας. Έχουμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλάζει ο κόσμο πολύ γρήγορα. Η συζήτηση για τα θέματα ηθικής είναι περισσότερο σημαντικό από ότι η συζήτηση την οικονομία. Και πρέπει να βρούμε κοινό τόπο συνεννόηση στην Ευρώπη με όλου σα. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή την ε, συνάντηση και για μία ακόμη φορά θέλω να σας πω ότι θα στηρίξει πλήρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει πλήρω αυτά που κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως αυτά που κάνει την πρόεδρο Μαγκίνε για αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you, Vice Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, και καλό ταξίδι, επειδή θα φύγετε. Πάντως, ε, θα ήθελα να εξηγήσω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε δύο πάνελ. Το πρώτο πάνελ αφορά το ε, μη χρησιμοποιημένο δυναμικό του τρέχοντος ε, νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε κατά πόσο χρειάζονται αλλαγές. Οπότε θα ήθελα να δώσω την ευθύνη και προεδρία του πρώτου πάνελ στη φίλη ε, Ντανούτα Χούμπνερ που είναι ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Ζητημάτων. Είναι εμπειρογνώμων σε αυτά τα θέματα, οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλά χέρια. Χαιρετούμε και τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρέπει να σας πω ότι δεν μας συμβαίνει πολύ συχνά εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορούμε να περάσουμε ένα ολόκληρο απόγευμα συζητώντας ένα θέμα το οποίο δεν είναι το Brexit. Ε, φαντάζομαι ότι και άλλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου ως προς αυτό. Είμαι επίσης πεπισμένη ότι όταν σκεφτόσασταν τι θα πείτε σήμερα το απόγευμα, ε, θα σκεφτήκατε και τον Ζακ Ντελόρ πριν από 25 χρόνια ξεκίνησε αυτόν τον διάλογο και ε, αναζήτησα και εγώ αυτό που είπε τότε, είπε ότι δεν θα επιτύχουμε στην Ευρώπη και αυτό στο πλαίσιο της συνθήκης του Μάστριχτ, είχε πει ότι δεν θα επιτύχουμε παρά μόνον δώσουμε ε, στην Ευρώπη, στην, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, μια, μια διανοητική ε, και πνευματική διάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Ζακ Ντελόρ πριν από 25 χρόνια είπε και θα μπορούσε να ισχύει και σήμερα. Χαίρομαι λοιπόν όλος ιδιαίτερος που σήμερα μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων γιατί σήμερα χρειάζεται αυτή την ηθική υποστήριξη Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται ε, να αφιερωθούμε στις αξίες μας και σε στενότερους δεσμούς με τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει επίσης να πω πολύ καθαρά ότι η Ευρώπη πάντοτε ε, ήταν συνειφασμένη με την αλλαγή ε, ακόμη και μέσω μεγάλων κρίσεων ε, μια έκκληση για αλλαγή σήμερα και η προσδοκία της αλλαγής μπορεί να, ε, γίνεται, να γίνει αισθητή σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα. Η ανάγκη για την αλλαγή στην Ευρώπη ήταν πάντοτε κάτι που απαιτεί το λόγο της πραγματικότητας γύρω μας και λόγω των ε, αξιών ε, που συναποτελούν την Ευρώπη, ε, αυτό είναι το ιδιαίτερο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όμως πάντοτε έχουμε κάποιες κοινέ αξίες, αυτές οι αξίες που ενέπνευσαν τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι, οποίοι, οι οποίες εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωμένες. Όμως τίθενται να αμφιβόλω σήμερα και όταν χάζον, χάνονται οι αξίες αυτές, ε, είμαστε κι εμείς χαμένοι. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αλλαγές ε, στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λόγω ανταπόκρισης ε, σε προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, ανάγκη για αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα που μερικές φορές ήρθαν με πολύ μικρά βήματα αλλά άλλες φορές από μεγάλες αλλαγές, αναθεωρήσεις και τους χάρτες πορείας που είναι η δίκευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο βαθιά ένα πιο βαθύ στοχασμό, γιατί είναι δύσκολες ε, οι ε, συνθήκες που αντιμετωπίσουμε σήμερα. Μπορούμε να ακούσουμε ότι συζητούμε πολλά, μπορούμε να πούμε ότι συζητούμε πολλά θέματα, την ξενοφοβία, ε, τον εθνικισμό, για ποιο λόγο αυτά τα φαινόμενα υπονομεύουν τη δημοκρατία και την νομιμότητα της Ευρώπης ε, η δημοκρατία που πρέπει να λειτουργεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είναι κάτι το οποίο τίθεται να αμφιβόλο. Το βλέπουμε και σε πολλές κυβερνήσεις και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές φορές ε, γίνεται παρέκκληση του κράτους δικαίου. Βλέπουμε μερικές φορές υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μεταξύ εθνικών ταυτοτήτων σε κράτη-μέλη και οι εκλογές μερικές φορές δεν είναι επαρκή ε, για να ε, εξασφαλίσουν τη δημοκρατία όταν υπάρχει μια έλλειψη δημοκρατικής κουλτούρας υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ε, ανεκτικότητας, βλέπουμε κατάρρευση παραδοσιακών ιδεοδών, βλέπουμε έναν πάρα πολύ καλό, κακό τρόπο πολιτικής ε, και βλέπουμε επίσης και πολύ επιδέξιους ε, πολιτικούς, όχι μόνο τους ε, δημαγωγούς που δημιουργούν όλες αυτές τις αντιευρωπαϊκές διαδικασίες και βλέπουμε πολύ κόσμο να αντιτίθεται πλέον στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν έναν, ένα κίνδυνο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον εθνικισμό πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να μας πάει προς τα πίσω. Υπάρχει μια μεγάλη απειλή στο μέλλον ε, της ε, Ευρώπης και αυτός είναι ο εθνικισμός όταν ε, θελήσαμε να, να... κάνουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου ε, Πολέμου, το κάναμε με βάση κάποιες αξίες οικουμενικές για την Ευρώπη, ε, όμως κάτι τέτοιο άρχισε να χάνεται με τις νέες γενναίες ε, και ε, δυστυχώς και με κάποιες ε, νέες γενναίες Ευρωπαίων ηγετών και παρά το γεγονός όσο ότι υπάρχει μια ενότητα εναντί στο Brexit αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ακόμη πολιτικού ηγέτε που θέλουν ε, να πάνε προ τα πίσω την ε, ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη πάντοτε ήταν ε, η Ευρώπη των πολιτών και για τους πολίτες. Όμως οι πολίτες σήμερα είναι πολύ διαφορετικοί από το πώς ήταν πριν από 60 ή 10 χρόνια καν και πρέπει να βρούμε διαφορετικούς τρόπους και μέσα να κερδίσουμε την δημόσια υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, την αλληλεγγύη, δύο βασικές θεμελιώδεις αξίες που έχουν χαθεί. Και εγώ έρχομαι από την Πολωνία, ένα, μια χώρα όπου οι πολίτες ε, απέρριψαν την πραγματικότητα χωρίς ελευθερία και αποφάσισαν μέσω δημοψηφίσματος ε, να είναι, ε, να είναι ε, τμήμα της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν ήταν πάντοτε τέλεια, έχουμε κάνει πολλά λάθη, το γνωρίζουμε αυτό και ο κατάλογος είναι μακρύς. όμως αυτά τα συλλογικά σφάλματα ε, χρήζουν σήμερα συλλογικής δράσης και εμείς ε, ως Ευρωπαίοι έχουμε ισχυρά δεμέλια για να ε, υπάρξει και πάλι ενότητα, οι επιστήμες, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, ε, αυτό το οποίο εκπροσωπείτε εσείς σήμερα, όλες τις αξίες που μοιραζόμαστε, που μας είναι κοινέ, χρειαζόμαστε και ηθική και αλληλεγγύη και θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σύντομή μου παρέμβαση λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και οι πολίτες και τα κράτη τα οποία ε, συνεργάζονται αλλά δεν ε, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να αρχίσει η συζήτηση και θα ήθελα να καλέσω τον Αρχιεπίσκοπο Ζων Κλοντ Χόλεριχ που ε, προέρχεται από την Καθολική Αρχιεπισκοπή του Λουξεμβούργου. Από το 2011 ε, είσαι στην Κομέσε, τη διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, ε, έκανα μάθημα ε, ευρωπαϊκών σπουδών στο ε, Πανεπιστήμιο Σόφια στο Τόκιο και για τους Ιάπωνες φοιτητές μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουν το περίπλοκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι ούτε ένα ενίο κράτος, αλλά ούτε και ένα είδος ε, ε, Ευρωπαϊκών ε, Ηνωμένων Εθνών. Κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία διολίσθηση. Το διακυβερνητικό γίνεται πιο ισχυρό και το κοινοτικό γίνεται πιο ασθενές. Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες, να καταλήξουμε σε ειδική πλειοψηφία ε, ή ακόμη περισσότερες δυσκολίες ε, ομοφωνίας με μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών. Μη με παρεξηγείτε, χαίρομαι για τον υψηλό αριθμό των κρατών μελών, όμως για να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων πρέπει ε, η κοινοτική διάσταση να καταστεί ισχυρότερη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν συχνά ε, την εικόνα ε, συγκρούσεων όσον αφορά το διακυβερνητικό επίπεδο και δίνουν ε, την εικόνα μιας διαιρεμένης Ευρώπης. Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει αν υπάρχουν εκλογές από εδώ και από εκεί και δεν υπάρχει καμία μετακίνηση σε επίπεδο διακυβερνητικό. Επίσης, ο ευρωσκεπτικισμός ε, ενδυναμώνεται έτσι και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να καταλάβουν τη χρησιμότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος της περιαγωγής ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άρχισε να ισχύει αυτό το μήνα είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απλοποιήσει τη ζωή των πολιτών της. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό ε, έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αποδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των ελίτ, αλλά όχι στη βάση ε, των πολιτών μας. Και αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημάδι, γιατί μπορεί να χάσουμε την δημοκρατική μας νομιμότητα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις υποψίες και να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μην ε, υπάρχει αμφιβολία ε, στο μυαλό και στις καρδιές των Ευρωπαίων πολιτών ότι η πολιτική τους ε, βούληση δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημοσίου χώρου ώστε τα στοιχεία της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης να γίνονται απολύτως αντιληπτά γιατί το ότι δεν υπάρχει τέτοιου ίδιου ε, δημόσιο χώρο ε, δίνει μια γραφειοκρατική εντύπωση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εντύπωση ενός διακυβερνητικού μακεβελισμού. Δεν λέω ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά αυτή την εντύπωση δίνουμε προς τα έξω. Και αυτό ε, έχει να ε, κάνει βέβαια και με τα συμφέροντα της, ε, της πολιτικής ελιτική, ελίτ και πολλές φορές αυτός, αυτή η έλλειψη του δημοσίου χώρου δημιουργεί προβλήματα στην θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες. Στο παρελθόν έχουμε δει ε, ότι ε, το να ληφθεί υπόψη πολιτική βούληση των πολιτών ε, είχε ως αποτέλεσμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το όνειρο είναι πάντοτε κάτι το πολύ γενικό. Κανένας δεν θυμάται τις λεπτομέρειες ενός όνειρου. Όμως το ευρωπαϊκό όνειρο έγινε μέσω λεπτομεριών πολλών συνθήκων που μερικές φορές τώρα δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε πια το όνειρο. Πρέπει λοιπόν να ξαναβρούμε αυτό το ευρωπαϊκό Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί καλύτερα να λύσει τα προβλήματα σήμερα και αύριο από, από ότι το κράτος μέλος μόνο του. Ας πάρουμε για παράδειγμα ε, το θέμα των προσφύγων. Ε, δεν θα σας κάνει εντύπωση ότι εγώ ως επίσκοπος ε, φυσικά μπορώ να ενθαρρύνω την αποδοχή των, και την υποδοχή των προσφύγων στα κράτη-μέλη. Ο, η, ο ανθρωπισμός, ο χριστιανικός το απαιτεί, όμως ας δούμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, μια, έναν ασαφή φόβο μεταξύ των Ευρωπαίων ε, αν η ροή των προσφύγων, των προσφύγων δεν σταματήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε με όλα τις τα μέσα να έχει μια πολιτική αλληλεγγύης ε, προς τις χώρες ε, στις οποίες πηγαίνουν οι πρόσφυγες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη δική τους σωματική ακεραιότητα αλλά και αυτή των παιδιών τους. Έχουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη και ότι δεν είναι παρούσα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα είδους σχέδιο Marshall για τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ώστε η εισρωή ε, των ε, οικονομικών μεταναστών να σταματήσει ε, δεν θα ήταν καλύτερο και για την Ευρώπη να είναι πιο ανεπτυγμένη η Αφρική. Προφανώς υπάρχουν πολλά μέτρα που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως υπάρχει αυτή ε, η διάκριση μεταξύ ενός μεγάλου εγχειρήματο που μπορεί να στεφθεί με επιτυχία και των μικρών λεπτομεριών που ε, είναι καλές αλλά δεν πείθουν τον κόσμο. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως σε επίπεδο ονείρου. Δώστε μας πάλι πίσω το ευρωπαϊκό όνειρο ένα όνειρο το οποίο προκύπτει από μία ε, ε Ιουδαϊκή και, ε, και χριστιανική παράδοση να ξαναπάρουμε και εμείς πάλι στα χέρια μας ε, το ευρωπαϊκό όνειρο χρησιμοποιώντας όλο το δυναμικό των συνθήκων για να μπορέσει ολόκληρη η δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθεί. Νομίζω ότι γι' αυτό διψάνε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατη, και ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι αναφερθήκατε σε αυτό ακριβώ το μεγάλο πρόβλημα που εγκυμο... και τον κίνδυνο που εγκυμονεί όταν όλο και περισσότερο πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση του διακυβερνητισμού στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζητήματα που προφανώς συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην επίσκοπο Ήρια Άσκολα, η εκτός από επίσκοπος του Ελσίνκη είναι επίσης ποιήτρια και είναι μεγάλη τιμή για μα που έχουμε μεταξύ των προσκεκλημένων και μια γυναίκα. Έχετε τον λόγο. Κυρία Άσκολα. Σας ευχαριστώ κυρία Συντονίστρια, κυρία Αντιπρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να εκφράσω ε, την χαρά και την, την ε, ε, ευχαρίστηση που μου δίνει το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυναντηθούμε μετά από ε, μόλις μισό χρόνο. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, των εκκλησιών και ημών του Κοινοβουλίου. Κατά την άποψή μου, όταν μια εκκλησία εμπλέκεται στη, σε τέτοιου τύπου συζητήσεις, σε τέτοιου τύπου διαλόγου, υπάρχουν δύο πειρασμοί Χαίρομαι βεβαίω που υπάρχει αυτή η εμπλοκή και αυτή η συμμετοχή των εκκλησιών. Όμω ποιοι είναι οι δύο πειρασμοί. Είτε η εκκλησία συμμετέχει με τρόπο πολύ επιφυλακτικό, είτε με τρόπο υπεροπτικό. Και ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό και ούτε πρόκειται να μας οδηγήσει σε σωστές λύσεις. Και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο περισσότερο σε βάθος αυτό το θέμα με βάση την δική μου εμπειρία. Κατάγομαι από τη Φιλανδία. Φέτος η Φιλανδία θα εορτάσει τα 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Θα θυμηθούμε, δεν θα ξεχάσουμε κατά τη διάρκεια αυτών των εορτασμών ότι μόλις 99 χρόνια πριν η Φινλανδία ε, σπαραζόταν από έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Και μόλις 150 χρόνια πριν, μικρό στην, ε, στη συγχρονική περίοδο αυτή, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν από την πείνα. Επομένως πρέπει να σκεφτούμε τι έγινε, πώς θα κατάφερε η Φινλανδία μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να γίνει μία από τις πλουσιότερες. Βασιστήκαμε στο θάρρος με το οποίο η ιδρυτέ του φιλανδικού, σύγχρονου φιλανδικού κράτους βασίστηκαν στην παροχή δωρεάν εκπαίδευση σε όλους. Οι προγονεί μα αποφάσισαν επίσης ότι σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στα σχολεία, θα έπρεπε να δίνει το δωρεάν συσίτιο. Αυτό παλαιότερα λειτουργήσε και ως κίνητρο ε, για τους γονείς για να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πέραν από το γεγονό ότι τα παιδιά θα μάθουν γραφική ανάγνωση. Και ιδιαίτερα τα κορίτσια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο αλφαβητισμός, τον γνωρίζει κανείς γραφή και ανάγνωση, είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή του στα κοινά, ανεξαρτήτως από την οικονομική ή κοινωνική κατάσταση των γονέων του. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, την λουθυρανική, αντιλαμβάνομαι την εκπαίδευση ως το κλειδί για να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη Ευρώπη. Να δώσουμε δηλαδή σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να μορφωθεί και φυσικά η εκπαίδευση δεν είναι μόνο οι γνώσεις, είναι και πολλά περισσότερα. Οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές κοινότητες γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήματα της εκπαίδευσης και έχουν εμπειρία ιδιαίτερα και με εκείνα τα παιδιά που δεν είχαν εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά μέσω της υποστήριξης που έλαβαν στο πλαίσιο ε, της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπόρεσαν να αποκτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία. Δεύτερον, όταν ακούω τη λέξη Ευρώπη, αντιλαμβάνομαι ότι έχει διαφορετική σημασία για διαφορετικούς ανθρώπους. Αναρωτιέμαι λοιπόν, υπάρχει κάποια κοινή ε, αντίληψη για την Ευρώπη, πόσο ενω, ενωμένη ε, είναι ή μπορεί να είναι δεδομένη τη ε, σημερινή κατάσταση. Για εμένα η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα στι Βρυξέλλε ή το Στρασβούργο. Για εμένα η Ευρώπη δεν ε, είναι μόνο αυτή η Ήπειρος που κατοικείται από ευτυχισμένους πλούσιους ανθρώπους. Είναι μια Ήπειρος στην οποία έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται από τη φτώχεια, από την ανεργία, που να ζουν υπό συνθήκες φόβου και στις εκκλησίες μας, στις θρησκευτικέ μας κοινότητες, τους ακούμε αυτούς τους ανθρώπους πολύ συχνά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν πολύ συχνά πρακτικές ιδέες, για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες μας. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν διάλογο, μια συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε οι ιδέες τους να μας εμπνεύσουν. Τρίτον, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να έχει ένα ξεκάθαρο όρομα όσον αφορά την κοινωνική εισόδα και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Αυτό ισχύει για όλους και για τα θεσμικά όργανα και για τις εκκλησίες. Σε αυτά τα ζητήματα χρειάζονται αποφάσεις. Αλλά επίσης χρειάζεται και ε, κάθε φορά μια ιστορία, ένα αφήγημα που θα εμπνεύσει. Τέταρτον, κατά την άποψή μου η Ευρώπη δεν είναι ένα νησί απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο που χτίζει φράχτες και προσπαθεί να περιχαρακωθεί. Η Ευρώπη αποτελεί μέρος των παγκοσμίων προκλήσεων, εξελίξεων και προσπαθεί να συμμετάσχει σε αυτές, δείχνοντας αλληλεγγύη απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της ανθρωπότητας. Εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, οι θρησκευτικές κοινότητες, οι εκκλησίες, μέσω των Ιεραποστολών, έχουν επαφές με απομακρυσμένα χωριά ε, και ανθρώπους που ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτές τις ε, ε, ιστορίες που φέρνουμε για τη δική μας συζήτηση, για τις δικές μας αποφάσεις. Πέμπτον, κατά την άποψή μου η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν καταφέρνει να αφουγκράζεται επαρκώς τους ε, εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι. Και μιλώ για όλους. Ένας άνεργος, μια ιερόδουλη από την Ανατολική Ευρώπη, ένας πανεπιστημιακός ο οποίος εκπέμπει ε, αρατσιστικό λόγο. Όλοι αυτοί έχουν κάτι να πούν σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να μεταβούμε από την εχθρότητα προς την αγάπη προς το πλησίον, προς τη φιλοξενία. Πιστεύω ότι όλες οι θρησκευτικές κοινότητες, όλες οι θρησκείες μπορούν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στην Ευρώπη από κοινού. Μια Ευρώπη όμως η οποία πρέπει να είναι ασφαλής, δίκαιη και πολυπολιτισμική. Να μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να γνωρίσει ο ένα τον άλλον καλύτερα. Και ιδιαίτερα να γνωρίσουμε ανθρώπους που διαφέρουν από εμάς. Να γνωρίσουμε τις παραδόσεις τους, τις εμπειρίες τους, τους φόβους τους και τα όνειρά τους. Κλείνω λοιπόν επιμένοντας στο ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι αγάπη, αγάπη το πλησίον, περιέργεια και αυτοπεποίθηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την Ευρώπη, σας. Προχωράμε στον καθηγητή του κ. Παντελή Καλαϊτζίδη από την Ελλάδα, διευθυντής του Πανεπιστημίου της, ε, του Βόλου για τις κοινωνικές μελέτες και έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Το μικρόφωνο σας παρακαλούμε. Το μικρόφωνο σας παρακαλούμε. Το μικρόφωνο σας. Uh, before starting... Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μου προς τον πρώτο αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μαγκίνες που μου προσεκάλεσε σε αυτή την ξέχουσα συνάντηση και στον το Χούτινεν, Γενικό Γραμματέα της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, της ΚΕΚ, που μου ανέθεσε να μιλήσω εκ μέρους της οργανώσεως αυτής σε αυτό τον πολύ σημαντικό διάλογο. Δεν είμαι ειδικό για τα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτε ειδικό για τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα διάφορα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ενομικά τις πολιτικές. Είμαι ένας Ορθόδοκος Χριστιανός Θεοθολόγος, ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, προερχόμενος από την χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή την Ελλάδα, μια χώρα η οποία είναι στην ε, αρνητική δημοσιότητα τώρα λόγω της φοβερής οικονομικής κρίσης ε, που περνά τα τελευταία 7 χρόνια. Θα προσεγγίσω μετά το κρίσιμο θέμα που συζητούμε από μια θεολογική έποψη και όχι από τεχνοκρατική ε, ή διαχειριστική, παιδιάς management. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα πρέπει να αποκαταστήσει τη δύναμή του και τη δυνατότητά του να θρίζει ανθρώπου από διάφορα υπόβαθρα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ξεπεράσει την κυριαρχούσα ιδέα που ήδη αναφέρθηκε Μία ενώσεως που καθορίζεται κυρίω από οικονομικού κανόνε ή μέτρα λιτότητα. Όπω δηλώθηκε στο έγγραφο ΚΕΚ με το θέμα ευημερία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, το ΚΕΚ, το έγγραφο της ΚΕΚ, εδώ και δεκαετίε η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σαν ένα όραμα, ένα εγχείρημα συμφιλίωσεω και ειρήνη. Αλλά μετά την υλοποίηση αυτή, βασική κινητήρια δύναμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία τη ήταν η επίτευξη στόχων που ε, ξεπερνούσαν την οικονομική συνεργασία. Αυτή η δήλωση λοιπόν που παρέθεσα μας υπενθυμίζει την Οικουμενική Χάρτα του 2001 και τη σχετική δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Και εδώ από τη Χάρτα Οικουμενικά αναφέρουμε ότι χωρίς κοινέ αξίες η ενότητα δεν μπορεί να διαρκέσει. Τέλος της παράθεσης από την Χάρτα Οικουμενικά. Οπότε ερχόμαστε στο πολύ κρίσιμο ερώτημα και θέμα των κοινών αξιών και το όραμα των ιδιωτικών πατέρων του Ευρωπαϊκού Ενώσεω ή των διακεκριμένων ηγετών, όπω ο πρώην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζακ Ντελόρ, που έλεγαν και παραθέτω τον κύριο Ντελόρ ότι δεν θα πετύχουμε με την Ευρώπη μόνο επί τη βάση νομικής τεχνογνωσίας ή οικονομικής ικανότητας. Αν δεν πετύχουμε δίνοντας μια ψυχή στην Ευρώπη τότε θα έχουμε αποτύχει. Τέλος τη παράθεση. Ένθερμα φρονώ ότι η παρούσα κρίση που αντιμετωπίζεται από την Ευρώπη είναι μια κρίση η οποία επωνόμευσε το ευρωπαϊκό εγχείρημα και το έκανε λιγότερο τακτικό για ανθρώπους εκτός και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετίζεται κατά πολύ με την έλλειψη ψυχής της Ευρώπης και επίσης σχετίζεται με την έλλειψη ελπίδας και οράματος. Και όταν η ψυχή της Ευρώπης και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον έχουν φύγει, με άλλα λόγια, όταν οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες όπως η ελευθερία, η λιλεγγύη, η δικαιοσύνη, το, το πώς θα ξεπεράσουμε τη φτώχεια και τον αποκλεισμό δεν ληφθούν υπόψη, τότε η ευημερία των στατιστικών στοιχείων αντικαθιστά την πραγματική ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε βαθμό να πιστεύετε ότι έχει ξεπεραστεί η κρίση και εδώ παραθέτω ότι η οικονομία έχει επιστρέψει στο μονοπάτι της ανάπτυξης και τα επίπεδα της ανεργίας μειώνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Λίγη παράθεση. Αυτό το αναφέρει και το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Αυτό διατείνεται το έγγραφο. Το ίδιο έγγραφο προβληματισμού δίνει 23% ποσοστά ανέργων για την Ισπανία και την Ελλάδα και περίπου 40% πάνω από 50% είναι στην πραγματικότητα για τους άνεργους νέους στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οποιουσδήποτε όμως επισκεφθεί την Αθήνα ή άλλη μεγάλη ελληνική πόλη, προσωπικά θα είναι μάρτυρας της ανθρωπιστικής καταστροφής που αντιμετωπίζει η χώρα μου τώρα για τα τελευταία 7 χρόνια και θα κατανοήσει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της ευημερία των στατιστικών στοιχείων και της πραγματικής ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Επίσης, όποιος είναι ευαίσθητος όσον αφορά τα μηνύματα που στέλνει ο λαός στην Ιταλία, την Ισπανία, έκομα και στη Γαλλία, και την αύξηση της επιρροής των δεξιών και αριστερών λαϊκιστικών κομμάτων σε αυτές τις χώρες, εκείνος ή εκείνοι δεν μπορούν παρά να αρχίσουν να διαρωτώνται όσον αφορά το έλλειμμα βασικών ευρωπαϊκών αξιών. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης χωρίς να συζητηθούν οι κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε απόπειρα να θεσπιστούν μέτρα για το ξεπέρασμα της παρούσης κρίσης. Θα πρέπει καταρχάς να κατανοήσουμε ποιες, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για την κρίση πριν αποφασίσουμε την ενδεδειγμένη θεραπεία. Επιτρέψτε μου εδώ να σας υπενθυμίσω ότι πέρα από τους, μεγάλους, τους πολλούς οικονομικούς λόγους που συχνά υπογραμμίζουν οι ειδικοί για το θέμα, θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε επί των ηθικών θεμάτων που σχετίζονται με τις πολιτικές για το χρέος, που συνδέονται άμεσα με την οικονομική και χρηματοστική κρίση και σχετίζεται επίσης με τη φτωχοποίηση μεγάλων τιμάτων του πληθυσμού στις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, τη μεγάλη αύξηση ανισοτήτων, την αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την εγκατάλειψη του ε, ε κράτους προνοίας. Δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε εμπειρογνώμων για τα χρηματοπιστωτικά. Και αν μιλώ σε αυτή την διάσκεψη, το κάνω αυτό μόνο υπό την ημοδιότητά μου σαν ένας χριστιανός διανοούμενος και σαν Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό, αυτή η ιδιότητα μου δίνει το δικαίωμα να αναφέρω την τρέχουσα κρίση που εξακολουθεί να ισχύει και να σοβεί στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν, συνεπώ, ότι είναι κατεπήγον να εξετάσουμε τι βασικέ επικρατούσε πολιτικέ στην Ευρώπη που όχι μόνο συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην περιθωριοποίηση μεγάλων κομματιών του πληθυσμού, αλλά επίσης οδηγούν σε ένα νέο διχασμό στην Ευρώπη. Διέρεση μεταξύ του Βορρά και του Νότου, που αντικαθιστά την παλιά διέρεση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σαν θεολόγος θα μπορούσα να, ε, να αναφερθώ σε πολλές βιβλικές ιστορίες και διηγήσεις από, το, από ε, Παλιά Διαθήκη, τη Νέα Διαθήκη, όσον αφορά το Ιωβιλαίο ε, την κρίση των κοινωνικών δικαιών την εκμετάλλευση των φτωχών και αδυνάμων κλπ. και τις κοινωνικές αδικίες. Όμως δεν θέλω να δημιουργήσω την εντύπωσή μου με τα επιχειρήματά μου, βιβλικές ιστορίες ή τα διάφορα κείμενα των πατέρων ότι προσφέρω ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί στην κοινωνία και στον τομέα του κοσμικού κράτους και των σχετικών πολιτικών. Γνωρίζω πλήρως ότι υπάρχει κοσμικός χαρακτήρας πλουραλιστικός της σύγχρονης, του σύγχρονου κράτους και υπάρχει εχθρότα ε, για διδασκαλική προσέγγιση από κριστικές αρχές. Εγώ δεν έχω κάποια, ε, δεν τρέφω αυτά πάντα στον αφορά τη μεταχριστιανική πραγματικότητα της σημερινής Ευρώπης. Εγώ ε, ενστερνίζομαι τον εσχατολογικό χαρακτήρα της Εκκλησίας και την απόσταση που υπάρχει από τις κοσμικές εξουσίες και τους θεσμούς. Και υποστηρίζω την αρχή ότι δεν μπορούμε τα βιβλικά κείμενα ή τις εντολές ε, του όρου των ελαιών, της όρου ομιλία, να τις κάνουμε αρχές που διέπουν ένα κράτος, διότι αυτό θα υπενθυμίζει θεοκρατία και ολοκληρωτισμό θρησκευτικό. Όμως, Πιστεύω ότι σαν χριστιανός θα μπορούσα να αναφερθώ στην βιβλική αξία της αλληλεγγύης που σημαίνει στην περίπτωσή μας το να υπερκεράσουμε τον συνολικό και εθνικό εγώ, ε, εγωισμό υπέρ ε, ενός ευρυτέρου σχήματος όπως είναι Ευρώπη. Εδώ και μερικά χρόνια, το 2013, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Γιούργεν Χάμπερμας σε μια μιλία του στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν με τίτλο «Δημοκρατία, αλληλεγγύη και ευρωπαϊκή κρίση» ζήτησε αλληλεγγύη σαν πολιτικό εγχείρημα ώστε να βγούμε από την κρίση η οποία καταστρέφει την Ευρώπη. Η συζήτηση όσον αφορά την αλληλεγγύη προβάλλει επίσης δύο άλλους θεολογικούς όρους. Διακονία, δηλαδή εξυπηρέτηση κοινότητας και όλων των συνανθρώπων και κοινωνία, δηλαδή κοινότητα, η πραγματική κοινωνία ή... Τέλος πάντων, δείχνει ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης, αν συζητούμε αυτές αρχές. Και παραθέτω το έγγραφο της ΚΕΚ. Σημαντικό κομμάτι της διακονίας συνεργάζεται με εκείνους που προσπαθεί να υπηρετεί. Αυτός ο ρόλος συμπεριλαμβάνει τον εντοπισμό ε, και την αντιμετώπιση των αδικιών σε κάθε επίπεδο, τοπικό, εθνικό και διεθνές. Σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες διαφορές εισοδήματος και πλούτου που χαρακτηρίζουν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Επίσης σημαίνει να προωθήσουμε ε, το σκοπό εκείνων και την προστασία εκείνων που αποκλείονται λόγω ε, φιλής, λόγω φίλου, λόγω θρησκείας, λόγω δυνατότητας ή λόγω ηλικίας. Πολλοί από τους Ορθόδοξους συναδέλφους α, ε, α, της Ευρώπης θεωρούν την Ευρώπη σαν κοινωνία και μια ενότητα στην διαφορά που θέλει να ε, έχουμε ε, ανοχή του άλλου και να δεχόμαστε και τη διαφορετικότητα, ούτω ώστε να πετύχουμε του στόχου του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό δεν ισχύει πάντα με εμά. Η άνευ οικονομική και χρηματοστική κρίση που περάσαμε τα τελευταία χρόνια, ίσω να δίνει την ευκαιρία στου λαού τη Νοτιού να μετανιώσουν και να κινηθούν επί πνευματικής, ηθικής και πολιτικής ορίμανσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αμφισβητηθούν και οι πολιτικές που εφαρμόζουν στους Ευρωπαίους ηγέτες και να εξεταστούν για να προσμετρήσουμε τις τραγικές και καταστροφικές συνέπειες που υπάρχουν όσον αφορά τους ανθρώπους, την κοινωνική ε, συνοχή και το μέλλον της Ευρώπης. Είναι κάτι που ε, δημιουργείται από τις νεοφιλελεύθερες ε, χρηματοστικές πολιτικές. Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης και παραθέτω τη Λευκή Βίβλο, κάθε φωνή θα πρέπει να εισακουστεί. Τέλος παράθεσης. Ελπίζω ότι η φωνή που τόλμησα να σηκώσω και τα κριτικά και αυτοκριτικά μου σχόλια συμβάλλουν ούτω ώστε να κατανοήσουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος πόσο ζωτικό είναι για την ίδια την Ευρώπη να παραμείνει για όλους μας δυτική, ανατολική, για τους δυτικούς ανατολικούς είναι ότι Ευρωπαίους ένα κοινό σπίτι και κοινή μοίρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, καθηγήτα ε, Καλαϊτζίδη, θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον αρχιραβίνο ε, των Βρυξελών, τον Αλμπέρ Γιγγί. Ε, που είναι επίση εκπρόσωπο της διάσκεψης ε, Ευρωπαίων Ραβίνων. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, η Ευρώπη η ιστορία της Ευρώπης ε, είναι 2.000 ετών και ήταν πάντοτε παράδοξη. Από τη μία ήταν ε, ε, γη υποδοχής, χειραφέτησης, ανάπτυξης, του Φρόιντ, του Αϊνστάιν και από την άλλη μία γη διωγμών, ε, γενοκτονιών, ε, πολέμων. Ε, έγινε η μεγαλύτερη γενοκτονία του κόσμου στο πλαίσιο μιας κοινωνίας πολιτισμένης και διαφωτισμένης. Νομίζω ότι σήμερα αποκτά συνείδηση η Ευρώπη πολλών προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η εβραϊκή κοινότητα και αναζητά θετικές λύσεις για τις ανησυχίες των μελών της κοινότητας αυτής και ε, έχω υπόψη μου κυρίως το πρόβλημα του αντισημιτισμού ε, στην Ευρώπη ε, της βίαιης τρομοκρατίας του σκοπό έχει να αποσταθεροποιήσει τις κοινότητές μας. Χάρη στη συνεχή δουλειά του κυρίου Ταγιάννη, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ε, του πρώτου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Τίμερμαν και της Αντιπροέδρου Μακίνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη σε μικρό χρονικό διάστημα έκανε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και ενέκρινε μία σειρά ε, μέτρων που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τις μειονότητές της. Θα ήθελα σήμερα να αποτίσω φόρο τιμής στους ανθρώπους αυτούς για όλη τη δουλειά που έχει γίνει και να τους συγχαρώ θερμά για ε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί γιατί ε, χάρη σε εκείνους ε, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκβάθους καρδίας. Όσον αφορά τώρα το μέλλον της Ευρώπης, θα ήθελα να εστιαστώ κατά κύριο λόγο σε δύο σημεία. Ε, την ολοκλήρωση και το, ε, το να ζούμε μαζί. Καταρχάς ε, πρέπει να υπενθυμίσουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της ολοκλήρωσης και της προσωμείωσης της αφομοίωσης. Ε, μπορούμε να ζούμε σε μία χώρα και να ε, συνεισφέρουμε με αρμονικό ε, τρόπο μέσω σεβασμού των θρησκευτικών πεπιθήσεων του καθενός και του, των νόμων του κράτους στο οποίο ζούμε. Αφομοίωση ουσιαστικά σημαίνει ότι χάνει κανείς την ιδιότητά του, την ταυτότητα του ε, για να γίνει ένα τμήμα της μάζας και να μην είναι πια ο εαυτός του. Σήμερα υπάρχει ένα ρεύμα, ένα ρεύμα επιμένω, ε, που θεωρεί ότι είναι, υπερέχει όλων των υπολείπων θρησκευτικών επεπιθύσεων ε, και θεωρεί ε, συνεπώς ότι είναι ο θεματοφύλακας της ουδετερότητας του κράτους. Για το ρεύμα αυτό πρέπει η θρησκεία πρέπει να είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα και δεν πρέπει να μπορεί να εκδηλώνεται ανοιχτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο και το οποίο μας ανησυχεί στο μέγιστο βαθμό. Στις 22 Μαΐου το Βαλονικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα διάταγμα που απο, απαγορεύει ε, τον ε, θρησκευτικό σφαγιασμό των ζώων. Στις 8 ε, Ιουλίου η φλαμανδική αυτοδιοίκηση θα κάνει το ίδιο και αυτό παρά την αρνητική τοποθέτηση του Συμβουλίου Επικρατείας. Οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι θα πρέπει λοιπόν να εισάγουν το κρέας από το εξωτερικό. Και αν γενικευθεί αυτό το μέτρο, ε, αυτό είναι το μέλλον των εβραϊκών κοινοτήτων και των μουσουλμανικών κοινοτήτων στο μέλλον, ε, γιατί αυτά θα ισχύσουν και για το μέλλον. Ε, αυτός ο νόμος είναι άδικος, γιατί έχουμε δώσει επιστημονικές, ε, επιστημονικά στοιχεία αναντήρητα, τα οποία λένε ότι δεν υποφέρουν περισσότερο ε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα ζώα. Για ποιο λόγο λοιπόν να επιτεθούμε στις θρησκευτικέ μειονότητες δεν ε, γίνεται δια της βίας, δεν είναι μέσω του φόβου και δεν είναι μέσω της καταστολής των πολιτιστικών διαφορών, μέσω της υποχρέωσης ε, των πολιτών ε, να δεχθούν κανόνες που θα οικοδομήσουμε το μέλλον της Ευρώπης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποιο είδους συνοχή. Πρέπει, είναι επιτακτικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους αν θέλουμε και οι άλλοι να μας σέβονται. Πρέπει να τιμούμε την ελευθερία των άλλων αν θέλουμε να τιμούν και εκείνοι τη δική μας ελευθερία. Η Ευρώπη χρειάζεται διάλογο με τις θρησκείες αν θέλει να αποφύγει στο έδαφος τους φονταμεταλισμό ε, κάθε είδους. Η Ευρώπη πρέπει να ε, ευνοήσει έναν ευρωπαϊκό Ιουδαϊσμό, ένα Ισλάμ ευρωπαϊκό που θα είναι σε θέση να εμπλουτίσουν τις αξίες και την κληρονομιά της αρνούμεθα μία Ευρώπη την οποία όπως έλεγε ο στρατηγός Ντεγκόλ που θα ήθελε να ε, συγχωνεύσει τους λαούς σαν ε, πουρέ από κάστανο. Ε, δεν λέμε ότι πρέπει να είναι απολύτως ομοιόμορφα όλα. Πρέπει να υπάρχει μια ενότητα χωρίς να ισοπεδώνεται η ταυτότητα και η ιδιαιτερότητα του καθενός, η ταυτότητα, η γλώσσα του, οι αξίες του, οι παραδόσεις του, η θρησκεία του μεταξύ του, της κοινωνικής ε, μεθόδου που θα ήταν ενδεχομένως επικίνδυνη ε, και την ε, κοσμικότητα, η οποία, την εκοσμίκευση η οποία θα μπορούσε να ισοπεδώσει τις διάφορες θρησκευτικέ πεπιθήσεις υπάρχει μία μέση οδός, μία τρίτη οδός, μία συμμαχία μεταξύ των θρησκευτικών αξιών και των δημοκρατικών αξιών. Ε, εδώ είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, εμείς ε, που οικοδομούμε την Ευρώπη του αύριο. Σε μια Ευρώπη ανταγωνισμού αυτή η συμμαχία θα έπρεπε να αποκαταστήσει τη γλώσσα της συνεργασίας. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ευθύνες και όχι μόνο στα δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι απαραίτητα, όμως οδηγούν σε συγκρούσεις που ε, τα δικαιώματα τα ίδια δεν μπορούν ε, να ε, επιλύσουν. Το δικαίωμα της γνώμης έναντι του δικαιώματος επιλογής, το δικαίωμα ελευθερίας ε, και δικαίωμα σεβασμού. Ε, τα δικαιώματα χωρίς ε, ευθύνες ε, είναι τα ενυπόθηκα δάνεια του μελλοντικού κόσμου. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα ακόμη σημείο το να, του να ζούμε μαζί μπορεί να σας σοκάρω. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλούμε για αυτό, για το για τη συνύπαρξη. Μπορώ να ζήσω, να συνυπάρξω εδώ και 40 ε, ε, χρόνια με τον γείτονά μου ε, που μένει απέναντι χωρίς να ξέρω ποιος είναι, χωρίς να ξέρω τι κάνει, χωρίς να ξέρω τι σκέφτεται και, παρα, και όμως συνυπάρχω μαζί του. Ζούμε μαζί. Αυτό, αυτόν τον όρο όμως πρέπει να το αλλάξουμε. Να μην λέμε συνύπαρξη, να λέμε ότι ε, δημιουργούμε κάτι μαζί. Όταν έχουμε κοινά εγχειρήματα και όταν μαζί ανταποκρινόμαστε σε μία πρόκληση, τότε ε, μπορούμε να καταλάβουμε ο άλλος ακριβώς πώς είναι. Είναι ένας εταίρος ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει, να βρω τη λύση ε, στο πρόβλημά μου. Δεν έχω ε, δεν τον φοβάμαι πια. Δεν είναι αντίπαλός μου. Αντιθέτως, ε, Ερχόμαστε πιο κοντά ένα στον άλλον. Ο Εμμανουέλ Λεβινάς ε, λέει ότι είναι αυτό η επιφύση του άλλου. Το να γνωρίζουμε τον άλλον όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι ναι, πρέπει να ευνοήσουμε την ε, καλύτερη γνώση του άλλου ε, μερικές φορές έχουμε μόνο προκαταλήψεις. Ε, είναι Εβραίος, ε, είναι ε, μουσουλμάνος, δεν ξέρουμε και πολλά για αυτούς. Οι γνώσεις μας συχνά περιορίζονται σε ψευδείς αλήθειες. Πρέπει να απαλείψουμε αυτές τις προκαταλήψεις. Πρέπει να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε και να εκτιμήσουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε αμοιβαία, αμοιβαίο σεβασμό στη διαφορά, δηλαδή να υπάρχει ενότητα εν μέσω πλουραλισμού. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που, που η Ευρώπη θα στέλνει στους πολίτες της. Κυρίες και κύριοι, ο Θεός μας έδωσε πολλές γλώσσες και πολλούς πολιτισμούς. Όμως, έναν μόνο κόσμο μέσα στον οποίο πρέπει να ζήσουμε. Και αυτός ο κόσμος συρρυκνώνεται μέρα με τη μέρα. Ε, θα μπορούσαμε εμείς, ε, οι χώρες και οι πολιτισμοί της Ευρώπης ε, με την τεράστια ένδοξη διαφορετικότητά τους να δημιουργήσουμε μια νέα συμμαχία για την Ευρώπη η οποία θα μπορέσει να διατηρήσει τις αξίες μας και τον πνευματικό μας πλούτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραβίνα Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο τελευταίο μέλος του πάνελ μας, τον κύριο Έλμα Μπροκ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας ε, Ευρωπαίος, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του για τις κοινέ αξίες που μας ενώνουν στην Ευρώπη. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Μπροκ θα έπρεπε να τον εφεύρουμε ήταν τόσο σημαντική η συνεισφορά του και στο Κοινοβούλιο αυτό και στην Ευρώπη γενικότερα. Κύριε κύριος Μπρόκοφ, σας ευχαριστώ Ντανούτα. Θα μιλήσω γερμανικά μιας και έχω τη δυνατότητα και μπορώ να εκφράσω και πολύ καλύτερα, να εκφραστώ πολύ καλύτερα για θρησκευτικού χαρακτήρα ζητήματα στην μετρική μου. Πάμε όμως στο δεύτερο άρθρο της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις ε, ε αξίες του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού των μειονοτήτων. Αυτές τις αξίες τις μοιράζονται όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία μαζί με την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανεξιθρησκεία, την αλληλεγγύη Και αυτά αναφέρονται και στη συνθήκη της Λισαβόνας και στο προήμιο της, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για αξίες οι οποίες βασίζονται στην κοινή πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Ευρώπης. Η πολιτική ομάδα η οποία την οποία εκπροσωπώ, θεωρεί και πάντοτε έχει υποστηρίξει ότι οι ευρωπαϊκές αξίες βασίζονται στην ιουδιακή χριστιανική παράδοση. Πρόκειται για πυλώνες της, ε, ε, των πολιτισμών που έχουμε στην Ήπειρό μας και ε, εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους σε τις χώρες μας. Με τις διαφορές τους. Στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι η πολυμορφία είναι, ήταν ε, και είναι μάλλον μια, ένα πλέον έκτημα. Το διαπιστώσαμε αυτό και το προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Εράσμου στην ε, που δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίζουν την ποικιλομορφία και τις, διαφορετικού τις διαφορετικούς πολιτισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να ξεπεράσει τις καταστροφές που, που προκάλεσε ο ναζισμός και ο κομμουνισμός. καταφέραμε να έχουμε 70 χρόνια ειρήνης στην Ήπειρό μας. Η Ευρώπη ε, είχε πολύ θετικέ επιπτώσεις, ε, ε, συνεισφορά μάλλον, σε όλα τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα νεοεισελθέντα κράτη-μέλη. της αξίας της ανεξιθρησκείας, του κράτους δικαίου Τη συμμεριζόμαστε όλοι. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να έχουμε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση. Προσωπικά είμαι καθολικός. Δεν θέλω όμως να ζω σε μια χώρα η οποία θα προσπαθήσει να επιβάλλει την καθολική πίστη στους πολίτες της. Και διαπιστώνω δυστυχώς ότι υπάρχουν μέχρι και μέλη της Εκκλησίας μου που δεν θα συμφωνούσαν μαζί μου σε αυτό το τελευταίο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι βαθύ πρόβλημα. Ε, που, πρέπει να μας προβληματίσει. Πώς δηλαδή θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια ανοιχτή κοινωνία με σεβασμό προς τον άλλο, χωρίς διακρίσεις και ε, με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ομαλές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, των διαφόρων πίστεων. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή, η επιδίωξη συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί το κράτος σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Το κράτος λαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους πολίτες. Και το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει αλλαγή των ε, πεπιθήσεων των πολιτών του. Είναι θέματα που έχουν αποσχολήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. εμεί πρόσφατα τα τελευταία χρόνια ε, συζητήσαμε το ζήτημα ε, της φαγή των ζώων ε, στη Γερμανία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα θέματος στο οποίο επισέρχεται το ζήτημα της θρησκείας, επίσης όμως τίθεται και το ζήτημα της ζωής των ζώων, της προστασίας των ζώων. Διαφορετικοί άνθρωποι λοιπόν θα προσλάβουν αυτόν τον δημοσιο διάλογο με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν κατατίζεται η νομοθεσία. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε νόμους τους οποίους τελικά να μην μπορούν να δεχθούν ε, μεγάλα μέρη της κοινωνίας μας όπως για παράδειγμα όλοι οι Εβραίοι ή όλοι οι Μουσουλμάνοι. Είναι απολύτως απαραίτητος λοιπόν ο σεβασμός της θρησκευτική πίστεως από την πλευρά των κρατών. Τα θέματα αυτά τα συζητούμε συχνά στο Κοινοβούλιο και εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Στοιχείο της ανεξιθρησκείας είναι η δυνατότητα να εκφράζει κανείς την άποψή του, να εκφράζει η ελευθερία της έκφρασης. Ε, για παράδειγμα, στη χώρα μου ε, ετέθη το ζήτημα του πώς μπορεί κανείς να εκφράζει θέσεις οι οποίες πιθανόν να θεωρούν προσβλητικές από τους μουσουλμάνους, ή από ορισμένους μουσουλμάνους ή από κάποια θρησκευτική κοινότητα. Όμως, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης με αυτή τη λογική. Η ανεξιθρησκεία σημαίνει ταυτόχρονα προστασία της ελευθερίας της έκφρασης έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να μπορεί να ακολουθεί τις θρησκευτικέ του πεπιθήσεις, να εκφράζει τις θρησκευτικέ του πεπιθήσεις, εφόσον αυτές δεν βλάπτουν κάποιον άλλον πολίτη. Η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου. Ε, ε, και είναι, πιστεύω, αναπόσπαστο στοιχείο της θρησκευτική ελευθερίας η δυνατότητα έκφρασης των θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεων οποιοδήποτε. Ε, σε μια, φυσικά με ειρηνικό τρόπο στο πλαίσιο ενός ε, ειρηνικού διαλόγου. Ανεξιθρησκεία δεν σημαίνει ότι η θρησκεία πρέπει να, να, παραγωνιστεί και να παραμένει μόνο στον ιδιωτικό, στην ιδιωτική σφαίρα και να μην έχει κάποιος τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του. κατά την άποψή μου και κατά την εμπειρία μου μάλιστα, είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσει κανείς με κάποιον μουσουλμάνο ε, όταν, έχει, όταν έχει, ε, γίνεται αυτή η συζήτηση επί την ε, βάση της ελευθερίας της έκφρασης, δηλαδή ότι και οι μεν και οι δε θα έχουν την δυνατότητα ανοιχτά να εκφράσουν τις πεπιθήσεις τους, τις θρησκευτικέ. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Πρέπει λοιπόν να είναι απολύτως ξεκάθαρα η σχέση μεταξύ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της θρησκευτική ελευθερίας, της ελευθερίας της έκφρασης. δυστυχώ ε, δυστυχώς παραδείγματα από κράτη-μέλη μάλιστα, στα οποία ε, έχει γίνει αυτό το λάθος όπου έχουμε πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο και μόνο επειδή έχουν την πλειοψηφία ε, μπορούν να λάβουν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να ε, υπονομεύουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων ή της μειοψηφίας. Ε, για παράδειγμα, τα τεκτενόμενα στην Πολωνία. Αν επιλέξουμε αυτόν τον δρόμο και πάλι θα χάσουμε την ελευθερία της έκφρασης και την, ελευθερία, και την, το σεβασμό στην διαφορετικότητα. Οι αξίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατυπώνονται στο άρθρο 2 που σας διάβασα στην αρχή της παρέμβασής μου θα πρέπει να είναι αυτές που μας καθοδηγούν. Εφόσον λοιπόν αποδεχόμαστε το κράτος δικαίου, η πλειοψηφία, η όποια πλειοψηφία, θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι δεν έχει, αυτό της δίνει το γεγονό ότι ε, διαθέτει την πλειοψηφία τη δυνατότητα να καταπιέσει μια μειονότητα, μια μειοψηφία. το ζήτημα αυτό αποτέλεσε κομβικής σημασία θέμα για την καθόλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για το ζήτημα της γλωσσικής πολυμορφίας, για παράδειγμα οι ιδρυτές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρωτεργάτες, ε, κατάγονταν όλοι από περιοχές ε, οι οποίες είχαν πληγεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αντιλαμβανόντουσαν την σημασία που έχει η προσπάθεια να υπερβούμε τα σύνορα. Δεν θεωρούσαν ότι το κράτος έθνος έχει πεθάνει, όμως καταλάβαιναν ότι το κράτος έθνος έχει τα όρια του και ότι χρειάζεται να τα υπερβούμε και να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρξει αλληλοκατανόηση μεταξύ των διαφορών κρατών. Αυτή η ιδέα είναι στην καρδιά της ύπαρξης ε, της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε ήταν απολύτως πρωτοποριακές αυτές οι ιδέες, όμως είναι αυτές ακριβώς οι οποίε μα προστάτευσαν επί τόσα χρόνια από την ανελευθερία, από τις δικτατορίε, για παράδειγμα, σε κάποιε χώρες. Χρειάστηκε λοιπόν να ξεπεράσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος και προσπαθήσαν οι πρωτεγάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα ώστε κανένα κράτος να μην ε, έχει τη δυνατότητα πλέον να πάει σε έναν πόλεμο παρόμοιο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Γι' αυτό ανησυχώ όταν βλέπω την άνοδο του εξτρεμισμού, του εθνικισμού όταν ακούω όλο και περισσότερες φωνές οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να βάλουμε το έθνος, το, το έθνος κράτος, το έθνος τους ε, πάνω από οτιδήποτε άλλο και πρέπει να αντιταχσόμαστε ε, σε αυτές τις ε, προσεγγίσεις, αυτές τις φωνές στο βαθμό που αποτελούν μια προσβολή των κοινών μας αξιών. Για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πίσω γυρίσουμε. Ε, δεν θα γυρίσουμε στο, στο, στο σκοτεινό μας παρελθόν. Βεβαίως χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ίδια συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται στη σημασία που έχει η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, η βελτίωση της ευημερία για όλους τους πολίτες, η προστασία του περιβάλλοντος ε, και η ενιαία αγορά αναφέρεται ως μέσο προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Πρόκειται λοιπόν για στόχους οι οποίοι είναι ήδη καταγεγραμμένοι και αναγνωρίζονται ως στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνθήκες της. Αυτό σημαίνει στην πράξη, στις, σε συγκεκριμένες πολιτικές, ότι πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως σας είπα, εξαιτίας εν μέρη ίσως και του υποβάθρου μου του προσωπικού, του γεγονός ότι είμαι καθολικός, Δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία στην αλληλεγγύη. Ε, με ενοχλεί όταν ακούω πολύ συχνά την επίκληση της επικουρικότητας στις ε, ευρωπαϊκές συζητήσεις. Ένα παράδειγμα. Ακούστηκε το ζήτημα της ενεργείας των νέων. Πώς σχετίζεται το ζήτημα της αλληλεγγύης με την ανεργία των νέων. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίδει περίπου 50 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ στις πλέον υποβαθμισμένε περιοχές, οικονομικά υποβαθμισμένε περιοχές. Αυτό είναι μια μορφή αλληλεγγύη. Θα μπορούσαμε βεβαίω να συζητήσουμε αν αυτό το ποσό πρέπει να, να αυξηθεί, να αλλάξουν τα κριτήρια με τα οποία ε, αποδίδεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά την εκλογή Μακρόν θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ζήτημα αυτό των διαρθρωτικών ταμείων που θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο. θυμάμαι ότι ακόμα και τις καλές εποχές, τις εποχές των, παλαι... των παχαίων Αγελάδων είχαμε 30% ανεργία των νέων κατά μέσο όρο. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 50%. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιλύσει το θέμα. Μπορεί όμως να επιληθεί σε εθνικό επίπεδο, όπως πιστεύω πως όχι. Κατά την άποψή μου, η ανεργία των νέων σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με την οικονομία της αγοράς. Ε, Γι' αυτό, αυτό που απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να έχουμε αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Πρωτίστως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Χρειάζεται λοιπόν μια διασύνδεση όλων αυτών. Το γενικό όφελος θα επιτευθεί αν κάθε πολίτης κάνει τη δουλειά του, το ΣΥΠΗΝ, για τον οικοκυριό, για το σπιτικό του. Όμως θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και για τους άλλους. Εγώ έτσι κατανοώ το χριστιανικό δόγμα και πάντα έτσι λειτουργούσα ω πολιτικό. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική φύση των ανθρώπων. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Υπάρχει κάποια ένταση και αν επιληθούν οι εντάσεις θα είναι προς το κοινό όφελος. Θα πρέπει αυτό να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα κομμάτι της συζητήσεως αφορά την επικουρικότητα, άλλο κομμάτι την αλληλεγγύη και πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά μαζί. Έτσι θα πετύχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλμερ. 12 λεπτά έχουμε για συζήτηση, ερωτήσεις. Όποιος επιθυμεί, ας μας το πει να λάβει το λόγο. Να υποβάλει ερώτηση ή να κάνει κάποιο σχόλιο. Ποιος είναι πρώτος, δεν γνωρίζω. Ποιος σήκωσε το χέρι πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. David Filton. Εκπροσωπώ την Αγγλικανική Εκκλησία και έχω κάποια σχόλια να κάνω. Εκ μέρους του Επισκόπου ε, κυρίου Έλλης που μας εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να αναφερθώ στο Brexit, δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό όλες, όλες, όλοι ψήφισαν να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, οι επισκοπές μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπερίσχυσε η Σοφία, δεν είχαμε σφιγμομετρήσει σωστά τον παλμό των ανθρώπων και ψήφισαν διαφορετικά. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Έκαναν, πήραν μια απόφαση ε, οι άνθρωποι και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά. Ένα τα θετικά λοιπόν του Brexit, όπως είπε και ο Κίβερ Χόφστατ, είναι ότι η αναχώρηση του Ευρωπαϊκού το Ηνωμένο Βασιλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως να οδηγήσει σε στενότερες σχέσεις μεταξύ των εναπομενών των κρατών μελών, των 27 στενότερες ε, σχέσεις οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν. Βλέπετε κάθε σκοτεινή πλευρά έχει και τη φωτεινή τη όψη. Μετά η Αγγλικανική Εκκλησία παραμένει πεπισμένη για τη σημασία ε, η ηθική στοιχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί ομιλητέ το ανέφεραν αυτό. Που βασίζεται στη συμφιλίωση και την ειρήνη. Να συναθρίζεται ο κόσμο, να συμφιλιώνεται ο κόσμο μεταξύ ε, των φοβερών εμπειριών ε, του πολέμου. Να προχωρήσουν μαζί τα κράτη για να λύσουν τα προβλήματά του ειρηνικά και όχι με την φωνή των όπλων. Όμω, δυστυχώ, καμία πλευρά στη συζήτηση του δημοψηφίσματο δεν το προέβαλε αυτό σωστά πέρσι, αυτό το επιχείρημα. Τρίτον, σαν Εκκλησία παραμένουμε άκρο ενδιαφερόμενοι και υποστηρίζουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αυτό διότι η Βρετανία θα έχει και πάλι και στο μέλλον σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι η μορφή αυτή τη ε, σχέση που θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Χιλιάδε Αγγλικανοί από όλο τον κόσμο ζουν εντό των κρατών μελών των 27 τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τρίτον, η Αγγλικανική Εκκλησία ε, βρίσκεται σε 167 χώρες και εκπροσωπείται και ενδιαφέρεται συνεχώς στην ε, ευόδοση του εγχειρήματο του ευρωπαϊκού όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη εξωτερικού εμπορίου, όλος ιδιαίτερος. Για το μέλλον, ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι να αναπτυχθεί, όχι μόνο σαν μια κοινή αγορά, αλλά σαν κοινωνική και πολιτική κοινότητα, εκεί όπου αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και η ευημερία όλων των ανθρώπων εκτιμούνται και προωθούνται. Τέλος, Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δεοντολογικές διαφορές και πολιτισμικές διαφορές στην Ευρώπη. Και ο καθηγητής από την Ελλάδα και άλλοι το ανέφεραν αυτόν, ότι αυτό θα πρέπει να καλυφθούν αν θέλουμε να γίνει πραγματική κοινότητα ανθρώπων και κρατών και εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Να πω όμα ότι πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε για την ε, δυνατότητα. Προτεστανική Εκκλησία της Γερμανίας, Κατρίν Χάτιγκερ, με λένε. Σε αυτά που είπε ο προλαλής σας, οι εκκλησίες πρέπει να μιλήσουν κατά του ε, εθνικισμού, αυτό που είπε και ο κύριος Μπροκ. Αυτό κάναμε τον Νοέμβριο, όταν η σύνοδός μας ε, συζήτησε ένα έγγραφο με τίτλο «Ευρώπη και αλληλεγγύη». Αυτό κάνουμε, αυτό συζητούμε οικουμενικές σχέσεις και ε, διαθρησκευτικός διάλογος πρέπει να ενισχυθούν για να ξεπεράσουμε τις διαφορές που βλέπουμε στην Ευρώπη. Μεγάλες διαφορές που είναι εμπόδια όσον αφορά το να ε, ομαδοποιήσουμε καλύτερα, να, να είναι πιο ενωμένη η Ευρώπη. Και θέλουμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Το Μάιο, στην ημέρα της Εκκλησίας, ε, οι κοσμικοί άνθρωποι ε, συναθρίστηκαν, 100.000 άνθρωποι στο Βερολίνο έγινε αυτή η Kirchen Tag και εκεί ε, είχαμε μια ημερίδα και το πάνελ συζήτησε σοβαρά το μέλος της, ομα... της Ευρώπης, συμμετείχε ο Επίτροπος Κισέτινγκ και ο κ. Μπρόκ εκεί. Και μέσω του διαλόγου μαζί σας με το Ευρωκοινοβούλιο και τις εκκλησίες και θρησκευτικού οργανισμούς θέλουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιακνουσάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γιακονσάρη. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Έχουμε τους διερμήνεις εδώ. Ευχαριστώ. Ο διάλογος, η συζήτηση ήταν βασικές λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν. Τα τόνισε αυτά τα στοιχεία και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Τίμερμανς. Τώρα είναι η εποχή να ακούμε, όπως είπε, εκείνους που διαφωνούν. Διότι Πολύ συζητήσαμε για τα προβλήματα του εξτρεμισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη, τα καταδικάζαμε τα φαινόμενα, δεν αναρωτηθήκαμε όμως γιατί συμβαίνουν αυτά, γιατί εξελίσσεται ούτως η κατάσταση. Πρέπει να συναντούμε τους άλλους ανθρώπους, να τους πλησιάζουμε. Το θέμα είναι με την τέταρτη αυτή βιομηχανική επανάσταση με την ε, τεχνολογία της πληροφορικής. Αυτή η τεχνολογία πώς επηρεάζει την κατάσταση. Γίνεται όλο και περισσότερη συζήτηση στο διαδίκτυο, Φερρυπίν. Όλο και περισσότερο συζητούμε όμως με ανθρώπους που συμφωνούν μαζί μας. Και αυτό οδηγεί και στο μίσος πολλές φορές. Και έχουμε και το φαινόμενο της οργής στα μέσα μαζικής δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης στη Φιλανδία και γίνεται μια φυσαλίδα που απομονώνεται από τους άλλους που σκέφτονται διαφορετικά. Δημιουργούνται ομάδες και εκεί μέσα στη μια φυσαλίδα κλιμακώνεται η οργή των συμφωνούντων. Θα πρέπει να συναντούνται και άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά. Να μην μένει ο καθένας στη φυσαλίδα τη δική του των κοινωνικών μέσων και του διαδικτύου. Να μην υπάρχει διαχωρισμός και να μην τροφοδοτείται έτσι η οργή και η μυσαλλοδοξία που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τώρα. Θα πρέπει να συναντούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους, να καθησυχάζονται οι φόβοι που δημιουργούνται, να μην δημιουργούνται από δύο πομπέοι τράγοι. Υπάρχει ισλαμοφοβία, αντισημιτισμός που αναπτύσσονται, παραδείγματο χάρη. Αυτά είναι φαινόμενα που υφίστανται δεν ωφελεί στο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτούς με τους οποίους δεν συμφωνούμε. Πρέπει να το συναντήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που απευθύνω προς όλους, εκκλησίες και πολιτικούς. Να συζητούμε με αυτούς που διαφωνούμε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Με ενέπνευσαν αυτά που άκουσα, αυτά που είπαν. Ήταν ε, ανανεωτικό μετά από αυτά που συζητούμε εδώ, που είναι οδηγίες, κανονισμοί κλπ. Ευχαριστώ. Τσάμπα Τσόγκα. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Όχι. Αν δεν υπάρχει άλλος, έχω μια ερώτηση από τους προσκεκλημένους μας και το πάνελ. Ερώτηση. Όπως τα βλέπετε εσείς και από την καθημερινή επικοινωνία σας με τον κόσμο. Κοινωνία πολιτών, διάφορους φορείς το αν αισθάνονται υπεύθυνοι οι άνθρωποι για την Ευρώπη. Είναι ζήτημα αυτό που το διαπιστώνουν αυτό να υφίσταται αυτό σαν πρόβλημα αυτοί με τους οποίους έχεις επαφή. Αν αισθάνονται υπεύθυνοι για την Ευρώπη οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλείτε. Ορίστε. Φοβούμαι. Θα μιλήσω και εγώ για το Brexit. Μετά το Brexit ο κόσμος έχει μεγαλύτερη επίγνωση το ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες στην Ευρώπη, να είμαστε αφοσιωμένοι. Αυτό διαπιστώνω από την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους της Εκκλησίας και εκπροσώπους ε, κοσμικών φορέων, τουλάχιστον στο Λουξεμβούργο. Από τη δική μου εμπειρία υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ γενεών και εντός των ε, δομών της Εκκλησίας. Η νεότερη γενιά θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ένα κομμάτι της καθημερινής τους ζωής μέσω της τεχνολογίας, ε, της πληροφορικής, ε, του ταξιδιού, προγράμματα, Σόκρατες κλπ. Αλλά στους μεγαλύτερους όταν ήρθα να έρθω στις Βρυξέλλες, χάρη, Κάποιο από του γυρότερου συναδέλφου μου είπαν Α, πάτε αύριο στην Ευρώπη. Μου λέει. Του λέω, είμαι ήδη στην Ευρώπη, τους λέω, του λέω. Α, πρέπει να προσέξουμε και τις εικόνες και τη ρητορική που χρησιμοποιούμε. Αυτό πιστεύω. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα αυτή τη φορά. Ε, Κυρία Πρόεδρε, στην τοποθέτησή σας, στην εισαγωγική, μιλήσατε για τον εθνικισμό στο σοβαρότερο πρόβλημα της Ευρώπης. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο από τι άλλα μέρη, από τις άλλες χώρες. Ε, κοντά σε όσα είπαν οι προλαλήσαντε, θα ήθελα να προσθέσω και αυτή τη διάσταση. Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν είναι πια δεδομένη, γιατί η κρίση την οποία δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει, τροφοδότησε τους επιμέρους εθνικισμούς, τροφοδότησε τα αισθήματα απογοήτευσης και απομάκρυνσης από το ευρωπαϊκό όραμα. Και επίση ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να θίξω στην εισήγησή μου γιατί ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος, αλλά το οποίο ήδη κάπου αναφέρθηκε είναι το θέμα ε, της προσφυγικής κρίσης και της μετανάστευσης. Ε, τα θέματα αυτά νομίζω ότι είναι σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησης και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας όταν προσπαθούμε να δούμε και να μιλήσουμε για το πόσο κοντά νιώθουν οι λαοί στο ευρωπαϊκό όρομα. Θα μου, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ακόμα μια διάσταση. Ε, προέρχομαι από μια χώρα, από την Ελλάδα, που θρησκευτικά ε, ανήκει στην σφαίρα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα, ένα, ακόμα μια πρόκληση ε, που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η πρόκληση αυτή ε, σχετίζεται με την υπέρβαση του παλαιού σχίσματος μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Χριστιανισμού. Οι, όσοι προερχόμαστε από ορθόδοξες χώρες έχουμε έντονο το αίσθημα ότι η παλιά αυτή διαίρεση δεν έχει ξεπεραστεί. Ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση νιώθουμε ως μια μειοψηφία. Αριθμητικά είμαστε μια, μια, μειοψηφία, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε μπορέσει απολύτως να ενταχτούμε στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι, στο κοινό ευρωπαϊκό όρομα. Και θα ευχόμαστε να υπάρξουν μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το πάνελ αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι η αποστολή εξετελέστη. Θα ήθελα όμως να πω κάτι ακόμη, γιατί νομίζω ότι Ακούσαμε πολλά καλά νέα για την Ευρώπη, για το δυναμικό της, τους κινδύνους, αλλά ακούσαμε και κάποια άσχημα νέα. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικός ο ρόλος ο παιδαγωγικός, γιατί οι εκκλησίες έχουν μεγάλη ευθύνη σε αυτό το τομέα και ξέρουμε ότι αν δεν συνεργαστούμε με τα παιδιά και τους νέους, να τους πούμε πώς μπορούν να ζουν ε, ε, σε μια κοινωνία με, διαφορετικότητα ε, δεν θα γίνει από μόνη της η Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τη διαμορφώνουμε και αυτό είναι κοινή μας ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του πρώτου πάνελ, ε, γιατί ήσασταν και πολύ λεπτομερείς και σεβαστήκατε τα χρονικά όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ε, επειδή εγώ όπως σας είπα απλώς ακούω σήμερα, ε, κατά κύριο λόγο, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε μια, ε, την Ευρώπη ώστε να είναι κατάλληλη για το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Mercedes Presso, η οποία θα προεδρεύσει. Είναι ε, για το μέλλον της Ευρώπης από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας δίνω τον έλεγχο για την Προεδρία του Πάνελ 2. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα μιλήσω στα γαλλικά, αν δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας. Αγαπητοί φίλοι και προσκεκλημένοι, είχα πει και ε, στο προηγούμενο πάνελ πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να ε, ανταποκριθεί σε πολλές ε, προκλήσεις, την προκλήσεις την άνοδο του εξτρεμισμού, την οικονομική κρίση, ε, την αύξηση των προσφύγων. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος και για μας νομίζω το μέσο, το εργαλείο που έχουμε κατά κύριο λόγο στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας του συνομοθέτη είναι ο διάλογος. Ο διάλογος ε, καταρχάς ε, ε, φυσικά με τους νομικούς εμπειρογνώμονες, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας αλλά και με την κοινωνία των πολιτών στην προκείμενη περίπτωση με τους εκπροσώπους των θρησκευτικών κοινοτήτων και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι είναι μία από τις κύριες και θεμελιώδεις αξίες ε, των συνθήκων μας επί των οποίων ε, εργαστήκαμε ως ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ε, την πρώτη έκθεση την διατυπώσαμε από κοινού με τον συνάδελφο Μπρόκ που μόλις έφυγε και προσπαθούμε να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν εντός των συνθήκων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο πλαίσιο μιας Ευρώπης πιο ισχυρής και πιο ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών Δεύτερη έκθεση του κυρίου Φερχόφστατ, ε, ο οποίος, ε, η οποία μάλιστα χρήζει περισσότερη συζήτηση ε, κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας και μέσω των υφισταμένων συνθήκων, αλλά και μέσω κάποιων αλλαγών που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, καλά επιθυμητά αποτελέσματα. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα της έκθεσης Φερχόφστατ γιατί νομίζω ότι έχει αναφερθεί ε, στο στο παρελθόν έχουν αναφερθεί τα περισσότερα, η σημασία της αύξησης ε, του βάρους της κοινοτικής μεθόδου. Η λειτουργία αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου των Υπουργών ε, είναι ε, κάτι το σχεδόν άγνωστο για τους πολίτες ε, και τις διάφορες ομάδες εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών. Ε, είναι ένα δεύτερο σώμα που ε, λειτουργεί με την ειδική πλειοψηφία. Θέλουμε όμως να είναι διαφανές, διαφανείς και σαφείς οι διαδικασίες. Με αλλαγή των συνθήκων θα μπορούσαμε μάλιστα η ορατότητα ε, να είναι μεγαλύτερη. Η ορατότητα του Συμβουλίου να είναι ένα είδος γερουσίας της Ευρώπης δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της ε, διαφορετικής, ε, διαφορετικού επίπεδου ε, ολοκλήρωσης, γιατί το κάθε κράτος μέλος είναι σε διαφορετικό επίπεδο, οπότε υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να κινηθούν με την ταχύτητα που θέλουν, άλλα κράτη-μέλη πιο γρήγορα, άλλα πιο αργά. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια που προσφάτως έχουν εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον, ε, το, την επιθυμία να ε, συμμετέχουν περισσότερο η ε, μεγαλύτερη επίσης δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης όπως και το ζήτημα των ιδίων πόρων το οποίο θα το γνωρίζετε. Αυτές είναι οι ιδέες λοιπόν τις οποίες μετέγραψε επί χάρτου κατά τους τελευταίους μήνες ε, η Επιτροπή μας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν επίσης. Ε, η ε, άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαδικασιών συμμετοχής ε, ε, μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικός. Αυτό έγινε από κοινού μεταξύ των Επιτροπών Συνταγματικών και Εξωτερικών Υποθέσεων. Μπορεί να φαίνεται αρκετά τεχνικό, αλλά όπως ε, υποθέτω ότι γνωρίζετε, και πολύ καλά μάλιστα, μερικές φορές αλλαγές μεγάλης σημασίας και ε, ευρύτατες πρέπει να γίνουν για να είναι πιο διαφανή ε, τα ευρωπαϊκά όργανα και πιο ικανά να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ε, πολιτών. Ειδικότερα ο διάλογος με τις ενώσεις και τις θρησκευτικές και μη θρησκευτικές κοινότητες, όπως ενθαρρύνεται στο πλαίσιο του άρθρου 17 της συνθήκης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο πλαίσιο της ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, ε, κοινωνιών ε, του πολίτη. Εσείς είστε, είστε εκείνη που ε, μεταφέρετε ε, τις απόψεις κοινωνίας των πολιτών σε εμάς και είστε και κοινωνοί ε, των αξιών αυτών προς τις κοινότητές σας. Θέλουμε δηλαδή όλα αυτά να τα θέσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο της δημιουργίας μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Κατα... γι' αυτό λοιπόν η άποψή σας μας είναι πολύτιμη και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πριν παρουσιάσω το δεύτερο πάνελ ε, που θα μπορούσε να είναι ο μύτος που συνδέει ε, όλες τις παρεμβάσεις σας. Φαίνεται να είναι μακριά όλα αυτά, αλλά είναι αύριο ουσιαστικά το ερώτημα που προκύπτει από το πάνελ αυτό είναι ποιες είναι οι, απο, ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ήρεμα τις προκλήσεις που μόλις ανέφερα και πολλές άλλες που ενδεχομένως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν ε, εξ ονόματος των θρησκευτικών κοινοτήτων και των κοινωνιών του πολίτη. Ε, να παρουσιάσω λοιπόν καταρχάς τον Εδεσιμότατο Χίλ, ο οποίος κάθεται εδώ δίπλα μου, πρόεδρος της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ο κύριος Χατζή, που είναι Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των, ε, ε, Ουλεμάδων του Μαρόκου, και ο επίσκοπος Ταμάς Φαμπινή από την Ευαγγελική Λουθυρανική Εκκλησία της Ουγγαρίας. Ε, έχουμε λοιπόν να ακούσουμε την άποψη και Ευρωπαίων αλλά και ε, φίλων μας ε, από την Μεσόγειο που είναι τμήμα και του παρελθόντος και του παρόντος και σίγουρα και του μέλλοντός μας. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για του πολύ 10 λεπτά ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και συζήτηση μετά. Λοιπόν, ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο εδεσιμότατος Κρίστοφερ Χίλ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω τις θέσεις που είναι και προσωπικές αλλά τι συμμερίζεται και η διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών η οποία εκπροσωπεί εκκλησίες που δεν βρίσκονται μόνο σε χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες χώρες όπως την Αρμενία και άλλες πολλές συμπεριλαμβανομένων και κρατών ε, τα οποία επιθυμούν κάποια στιγμή να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν εδώ στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ε, γιατί ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου ε, στικόμενος στο πόσο μπορεί να θεωρηθεί ηρωνία του γεγονό ότι ένας Βρετανός, όπως εγώ, έρχεται εδώ να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά έχω υποστηρίξει την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμουν από ε, του μέλου του 48%, όχι του 52%. Α, όχι μόνο η πολιτική, αλλά και θρησκευτικέ κοινότητε και ολόκληρε κοινότητε στη Βρετανία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συζητήσουν και να αντιληφθούν τι επιπτώσει σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητα, όπω πολύ καλά το γνωρίζετε εσεί εδώ. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρω να σας δώσω συγκεκριμένες και απλές ε, προτάσεις, συστάσεις για το ποια θα πρέπει να είναι οι αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στη συνθήκη της Λισαβόνης. Όχι. Νομίζω ότι ανταυτού θα ήταν πιο χρήσιμο να συζητήσουμε θέματα ε, που αφορούν στο όραμα, όχι τι λεπτομέρειε, Ότι αυτή είναι η αξία αυτή τη συζήτηση, αυτού του διαλόγου. Πιστεύω ότι η ενίσχυση του άρθρου 17 της συνθήκης της Λισαβόνας στο σημερινό, όπως προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, όπω ήδη αναφέρθηκε τον ε, καθηγητή κ. Καλατζήρη, η ε, διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών διατύπωσε ανέφερε την ε, σημασία των κοινών αξιών. Έγινε, αναφέρθηκε ήδη η παράθεση ότι χωρίς κοινέ αξίες δεν μπορούμε να επιτύχουμε την Ένωση. Και αναφέρθηκε ήδη η Οικουμενική Χάρτα, στην οποία οι χριστιανικές εκκλησίες της Ευρώπης δεσμεύτηκαν να συνεργάζονται προς μια Ευρώπη ε, κοινωνικά ευαίσθητη, ανθρωπιστική, στην οποία θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία και στην οποία θα κατησχύουν οι αξίες της συμμετοχής και του κράτους δικαίου, υπερβαίνοντας τα όρια των θρησκευτικών ή πολιτικών διαχωρισμών. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή διάγουμε μια περίοδο απογοήτευσης. Απογοήτευσης από την παγκοσμιοποίηση, απογοήτευση η πολιτικων διαχωρισμων δυστυχως βρισκει τη στιγμη διαγουμε εντείνεται από τις ε, ε, εντυνόμενες κοινωνικές ε, ανισότητες από την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και στην οποία διαπιστώνουμε μια άνοδο του λαϊκισμού, του εθνικισμού, ακόμα και του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, ε, της εχθρότητας κατά των μουσουλμάνων κτλ. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η απογοήτευση είναι ορατή και υπαρκτή και στο εσωτερικό των εκκλησιών. Ε, και οι εκκλησίες αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τα απογοητευμένα μέλη των κοινωνοτήτων τους, όπως ήδη αναφέρθηκε. Δεν μπορούμε να ζούμε σε γυάλινους πύργους. Για την ακρίβεια, για να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον ζούμε σε γυάλινους πύργους. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να ξανακατεύουμε στην, στη, στη, στη γη. Έχει υπάρχει ένα ρητό στα αγγλικά να μην πετά κανείς πέτρες όταν ζει σε μια γυάλινο πύργο. Ε, και εγώ θέλω να το πάω ένα βήμα παραπέρα, ο αναμάρτητος να ρίξει τον πρώτο λίθο. Η Ευρώπη έχει κάποια επιτεύγματα στα οποία θα πρέπει να ε, επιμείνουμε, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Από το 54 έχουμε τη συνθήκη για τα, κοινωνικά δικαιώματα, την χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το κοινό προϋπολογισμό. Και εδώ επιτρέψτε μου ένα πολιτικό σχόλιο να μην, γίνουν, να μην μεταφερθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αξιοποιούνταν ε, για ανθρωπιστικούς σκοπούς, να μην μεταφερθούν προς ζητήματα άμυνα, όσο σημαντική και να είναι η ασφάλεια. Είναι ιερό αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού. Αναφέρθηκαν πολλοί ομιλητέ ομιλητές στην ομιλία του Ζακ Τελόρ στους προσώπους των εκκλησιών. στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από τότε όμως έχουν αλλάξει πολλά. Όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολιόταν με ζητήματα οικονομικά και ζητήματα ανάπτυξης. Για, για εύλογους λόγους. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ιδίω μετά τις διευρύνσεις ήδη από τις πρώτες διευρύνσεις, μετά τα έξι μέλη, όλο και περισσότερο στεκόμασταν στα ζητήματα της, κοινής, της ενίας αγοράς, στα οικονομικά ζητήματα. Ήδη αυτό, ήδη αυτό ήταν ξεκάθαρο από το 7ο κράτος μέλος που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Και κάπως θα πρέπει να γυρίσουμε στα ζητήματα τα κοινωνικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, από τις κοινωνικές ανισότητες, από την τρομοκρατία, από τα προβλήματα ασφαλείας. Ε, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο σημαντικές και ουσιαστικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο χώρος Σέγγεν. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για την ΟΝΕ, ε, για την διακυβέρνηση του κοινού νομίσματος. Ε, αυτό είναι ευαίσθητο θέμα. Αναφέρθηκε ήδη το ζήτημα της ε, διάστασης μεταξύ της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας. Είναι κάτι ξεχωριστό η εθνική κυριαρχία από τον εθνικισμό. Είναι κάτι ξεχωριστό η αλληλεγγύη. Είναι κάτι ξεχωριστό η επικουρικότητα. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και πιστεύω ότι οι χριστιανικές εκκλησίες μπορούν να συνεισφέρουν στο διάλογο αυτό γιατί διαφορετικά οδηγούμαστε σε ένταση ενό προβλήματος που γνωρίζετε ήδη καλά, του δημοκρατικού ελλείμματο. Γιατί όπως θα ε, παρατηρήσατε και στο δημοψήφισμα της ε, Μεγάλης Βρετανίας, το ζήτημα δεν ήταν μόνο το θέμα της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, αλλά επίση υπήρχε και μια υποφόσκουσα συζήτηση η οποία επηρέασε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όσον αφορά την έλλειμμα δημοκρατία στο εσωτερικό του Ενωμένου Βασιλείου, της ε, αυξανόμενης εξουσία του Westminster σε σχέση με τι τοπικές κυβερνήσεις. Και έρχομαι στα τελευταία παρατήρηση που θα θέλω να κάνω στην διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών Όπω διατυπώνεται το αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση στο κείμενο που ανέφερε και ο καθηγητή Καλεντζίδης, αναφερθήκαμε στην έννοια του κοινού μα σπιτιού. Δεν σημαίνει ότι απλώ έχουμε γείτονε που δεν γνωρίζουμε. Είναι μια ιδέα βαθύτερη. Ε, ζούμε όλοι στο ίδιο σπίτι, σε, απλώς σε διαφορετικά δωμάτια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε και να δίνουμε ε, την ε, θέση που τους αναλογεί στις διαφορετικές, ε, στους διαφορετικούς πολιτισμούς, στις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον γαλλικό πολιτισμό, τον γερμανικό πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν προσπαθούμε να εξαλείψουμε αυτές τις διαφορές. Τέλος. το ερώτημα τι μπορούν να κάνουν οι εκκλησίες. Ο αντιπρόεδρος Τίμερμαντς ήδη είπε ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι περάσαμε πολλές, πολλούς αιώνες με πολέμους μεταξύ των εκκλησιών. Και σταδιακά με το ε, ε, οικουμενικό κίνημα περάσαμε από αυτές τις συγκρούσεις σε μια ε, προσπάθεια συνεργασίας και διαλόγου. Μέσω αυτής της διαδικασίας του οικονομικού κινήματος μάθαμε και εμείς στις εκκλησίες πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας και προσπαθούμε τώρα πλέον να απευθυνθούμε και σε άλλες ε, θρησκευτικέ κοινότητες πέραν των χριστιανικών, για παράδειγμα τους Εβραίους. Ε, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος με τις θρησκευτικές κοινότητες αυτές. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μια κάποια εμπειρία. Και καταφέρνουμε να κρατήσουμε την ουσιαστική συζήτηση χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα μιαν μιας βαρετών αναφορών στη συνθήκη της Λισαβόνας και γραφειοκρατικών προβλημάτων όπως συχνά γίνεται εδώ. Αυτή την προσέγγιση πιστεύω θα έπρεπε να ακολουθήσουμε και ε, στον διάλογο ε, εντός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη φοβάστε την συζήτηση, τον διάλογο με τις θρησκευτικέ κοινότητες. Οι εκκλησίες μας μετά από αιώνες συγκρούσεων κατάφεραν να βρουν μια κοινή γλώσσα και να συνεννοούνται και σιγά σιγά να ξεκινούν και μια συζήτηση με αλόθρησκους. Αυτό θέλουμε να συνεισφέρουμε στον διάλογο που προσπαθεί να ξεκινήσει και εντός της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή ευκαιρία που μου δίδεται και σε συναμική κοινότητα που διαβεί σε Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι κάτι σαν άσκηση, εναρμόνισης. του να πιστεύει κανείς σε κάτι και το να ανήκει. Του πιστεύει και το ανήκει. Αδιαφεσβήτητα, η Ευρώπη περνά μια περίοδο βεβαιότητας. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, δεν είναι εύκολο να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κυρίως ε, μετά από το Brexit, την προσφυγική κρίση και τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι νέες προκρίσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την ευημερία που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ε, οδηγεί στην αντιμετώπιση μιας αναλλακτική. Περισσότερη Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα της Ευρώπης ή νέα σύλληψη της ενίας, νέο όραμα για αύριο. Οι ευρωσκεπτικιστές επέμεναν πιστεύοντας ότι το Brexit μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εναπομένουσε χώρε αρπάζονται από την ελπίδα θα ξεπεράσουν την καταιγίδα οι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θα βγουν ισχυρότερε. Η ιδέα τη Ευρώπη στο κάτω-κάτω ε, είχε το, εμπεριέχει το όραμα του Αλτιέρο Σπινέλη και το Ερνέστο Ρώση που μας πέρασε μέσα από τις κακουχίες των δυσκολιών. Πολιτικοί κρατούμενοι που είχαν φυλακιστεί φασιστικά καθεστώτα κατά τη διάρκεια Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ζήσαμε. Το Brexit δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης, να αναδομήσουμε τους ε, θεσμούς, ούτως ώστε να, να αλλάξουμε την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν προθυμία επί τη ευκαιρία της 60ης επαιτίου των συνθήκων της Ρώμης έχουμε την ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεκινήσουμε προσπάθεια συμφωνίας για τις επόμενες δεκαετίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, το να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότητα και γρήγορα. Τέτοιου είδου εκφράσει. Η εξυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τέτοιε εκφράσεις δεν μπορούν να παραμείνουν παρατήρητες. Τι σημαίνει ο εξυγχρονισμός των σύγχρονων ευρωπαϊκών θεσμών. Να εξυγχρονίσουμε Σημαίνει τι, επιτάχυνση του ρυθμού της αλλαγής για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου κινείται με φρενήρις ρυθμούς. Επίσης χρειάζεται επικαιροποίηση, αναδιατύπωση, εξυγχρονισμός των δομών εξουσιών και λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ανώσεως. Όποιο και να ο ρυθμό τη μεταρρύθμιση, η μορφή τη μεταρρύθμιση, το όνειρο περισσότερο ενωμένη Ευρώπη δεν θα αναζωογονηθεί αν δεν υπάρχει αναζωογόνηση πνευματική φύσεω παραλίλω. Για επιτάχυνση τη αλλαγή και πολλαπλασιασμό των διαφόρων ενδεχομένων και σχεδίων, αυτά είναι προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουμε μόνο οι Ευρωπαίοι αλλά και όλοι οι άλλοι λαοί στον κόσμο. Ένα από του λόγου πίσω από την αύξηση του κενού μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των πολιτών αυτή είναι η αδυναμία μας σαν πολίτες να αντιμετωπίσουμε τον ταχαίως ε, μεταβαλλόμενο κόσμο και περιβάλλον. Και έτσι δεν μπορούμε να προβληματιστούμε και να βγάλουμε λογική από τις δράσεις μας. Ε, πολλό μάλλον δεν να σχεδιάσουμε μελλοντικέ δράσει. Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετάχυναν το, τη θεωρία του τέλου, Δηλαδή ενεργοποιείται ε, μια νέα ηθαγένεια άτακτη που έχει ισχύ μέσω των δικτύων αυτών. Ο νέος πολίτης όμως αναπτύσσει ε, νοοτροπίες που βασίζονται επί επιδικτικού χαρακτήρα, εγωιστικού χαρακτήρα. Άρα τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν. Χρειάζεται μια επανεφεύρεση της εσωτερική δυναμικής. Δύσκολο όμως. Και είναι δύσκολο να επιτεθεί και συνένεση για τη μελλοντική πρόοδο. Τα νέα κοινωνικής δικτύωσης έχουν απελευθερώσει τους πολίτες και μπορούν να πιέσουν τους εκπροσώπους δημοκρατία οι πολίτες, όμως αυτά τα μέσα μας οδήγησαν σε λαϊκισμό, εθνικισμό και αναρχικέ κοινωνίες χωρίς κατευθυντήριες αρχές. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση είναι ωφέλιμα. Απελευθερών τον άνθρωπο, ναι. Όμως υπάρχει πρόβλημα. Όταν η απελευθέρωση του πολίτη γίνεται αυτός σκοπός, δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτή ε, δεν θα οδηγήσει σε μείωση της κοινωνικής ολοκληρώσεως. Η κοινωνική ολοκλήρωση της Ευρώπης εμποδίζεται από την απελευθέρωση δυνάμεων και φορέων διάλυσης. Είναι μέσα απελευθέρωση τα δίκτυα αυτά. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση δεν μπορούν όμω να επανσυνδέσουν κοινότητε και να δημιουργήσουν δημόσιο χώρο ευρωπαϊκό για να αποφευθεί ο εθνικισμό εκτό αν κάποια εξωτερική αρχή φημώσει τι ευρωπαϊκέ φωνέ αυτές. Αυτό ακούγεται σαν ολοκληρωτική ε, όμως προπαγάνδα. Τώρα περισσότερο από ποτέ λοιπόν η Ευρώπη χρειάζεται διακαώ μια ψυχή. Αν και η ψυχή δίνει και μία συνεπάγεται και μία ε, αυτοπιθαρχία. Και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σαν να είναι μια πολύ γλυκιά θηλιά, δεσμός. Και λέει ότι η ελευθερία... Ε, η, ε, λοιπόν, οι γλυκές ελευθερίες μπορούν να ζουν μόνο αν υπάρχει ένας δεσμός, κάποια δεσμά τα οποία είναι γλυκά στη φύση τους. Καλούμε την, Ευρωπαίου τους Ευρωπαίους να ταπεινωθούν. Είναι ζωτική σημασία οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να συνεχίσουν επικοδομητικές προσπάθειες σε επαφή με προσώπους των θρησκειών. Όμως, είναι σαν να σπέρνουμε άγωνο χώμα. Αν πίσω από αυτή την προσπάθεια προδικάζουμε τον εξευρωπαϊσμό των θρησκειών ή να δώσουμε θρησκευτικό χαρακτήρα στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα ε, ταυτότητας και για το πόσο θρησκευτική είναι η Ευρώπη, να μην συζητάμε αυτά. Η θρησκεία πώς ορίζεται γεωγραφικά, αυτό δεν ταιριάζει με τι ανάγκε που έχει η Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της παγκοσμιοποίηση η Ευρώπη. Ε, ο ξεφορβαισμός του Ισλάμ, σαν απόπειρα, τι συνεπάγεται. Ε, ενίσχυση διαφόρων διαλεκτικών που οδηγούν σε κρίση και πολιτισμούς που δεν μπορούν να συντεριάξουν κλείσιμο και άνοιγμα. Η αιμονή επιμειώσεως ταυτότητας στη γεωγραφική διάσταση οδηγεί σε ταυτότητες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε ξένους πολιτισμούς, δικό μας πολιτισμό, δική μας κουλτούρα. Απ' την άλλη πλευρά του νομίσματος, αν θεωρούμε ότι η θρησκεία είναι ο μοναδικός σωτήρας, οδηγεί κάποιους εκπροσώπους της θρησκείας να δίνουν θρησκευτική ταυτότητα στην Ευρώπη. Και εφόσον όλες τις θρησκείες διατείνονται ότι μπορούν να σώσουν, η προσπάθεια να δώσουν μια θρησκευτική ταυτότητα στην Ευρώπη είναι κάτι θανάσιμο για την ευρωπαϊκή και θρησκευτική ποικιλομορφία. Άρα, πόσοι οι θρησκείες μπορούν να συμβάλλουν στο να δώσουν ψυχή στην Ευρώπη, αν δεν μπορούν αυτές να εκχριστιανίσουν, εξισλαμίσουν, εξιοδίσουν την Ευρώπη. Και πώς μπορεί να προχωρήσει το σκεφτικό εγχείρημα αν δεν εξευρωπαϊστούν οι θρησκείες. Μόνο μια λύση υπάρχει κοινή δράση δεν είναι το τι είμαστε ή πόσο Ευρωπαίοι είμαστε που πειράζει και νοιάζει και έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουμε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ύψη της σημασίας είναι οι συνεδριάσει υψηλού επίπεδου με κοσόπου των θρησκειών πρέπει να στιάζονται επί σχεδίων η κοινή δράση. Για τη διαφύλαξη της Ευρώπης σαν χώρου ισότητας, ποικιλομορφίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δώσουμε το παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια τρίτη παρέμβαση από τον επίσκοπο Ταμάς Φαμπινή. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς ε, τελευταίος, αλλά θα προσπαθήσω να μην σας κοιμήσω. Παρακαλώ όμως προσπαθήστε κι εσείς να μην αποκοιμηθείτε. Υπάρχει ένας μύθος και ένα όραμα για την Ευρώπη και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των δύο. Ο μύθος από την ελληνική μυθολογία είναι γνωστός. Ο Δίας, ε, ο αρχηγός των θεών, ε, ερωτεύτηκε την όμορφη πριγκίπισσα της Φινίκης στην Ευρώπη, μεταμορφώθηκε σε λευκό τάβρο, πήρε την πριγκίπισσα μαζί του ε, και την πήγε στην Κρήτη. Γεννήθηκαν τρία παιδιά και σύμφωνα με τον μύθο το όνομα της Υπήρου μας προέρχεται από την Ασιατική πριγκίπισσα. Εκτός από το μύθο όμως υπάρχει και ένα όρημα που μας οδηγεί πίσω στην Ασία. Όπως αναφέρεται στις βιβλικές πράξεις, κεφάλαιο 16, ένας Μακεδόν εμφανίστηκε στον Άγιο Παύλο ε, κατά τη διάρκεια της νύχτας και του είπε «Έλα να μας βοηθήσεις». Από ό,τι κατάλαβα, αυτό ήταν μια κραυγή για βοήθεια από την ε, ε, βέβηλη Ευρώπη προς τους Ιουδαίους και τον επερχόμενο χριστιανισμό. Ο Παύλος ανταποκρίθηκε σε αυτή την κραυγή βοήθειας και κήρυξε το Ευαγγέλιο και στην Ευρώπη, αναβιώνοντας το ήδη αποδυναμωμένο ελληνορωμαϊκό πλαίσιο. Και από αυτή τη δουλειά προέκυψε η Νέα Ευρώπη. Ε, αυτό μοιάζει με το όραμα ε, για το οποίο μίλησε προηγουμένως ο Αρχιεπίσκοπος του Λουξεμβούργου. Ε, με κάθε σεβασμό στους παλαιότερους αρχαίους πληθυσμούς, πιστεύω ότι πρέπει να εκπροσωπούμε σήμερα το όραμα και όχι το μύθο στην Ευρώπη. Σύμφωνα όμως με τις εμπειρίες μας και στη δυτική και στην ανατολική πλευρά της Υπήρου, η Ευρώπη φαίνεται να βυθίζεται σε μια παγανιστική, νεοπαγανιστική κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε δύο διακριτές μορφές αυτού του φαινομένου και θα είμαι μάλλον επιγραμματικός επειδή δεν έχω χρόνο. Στην Ευρώπη έχουμε, υπάρχει μια δραματική μείωση της επιρροής ε, του Ευαγγελίου ε, που ανανέωσε την Ήπειρό μας πριν από 2.000 χρόνια. Υπάρχουν και μερικά ε, συγκριτικά φαινόμενα. Το ανατολικό τμήμα της Ήπειρου ξεκίνησε από την αποπεριφερειοποίηση υπό την κομμουνιστική επιρροή και ακόμη και αν κάποιες ιστορίες ε, πίστης. Παράλληλα, η Δυτική, η Δύση άρχισε σιγά σιγά να εγκαταλείπει τα χριστιανικά οχυρά της και άρχισε να απομακρύνεται από ε, τον ε, επαναστατικό χαρακτήρα του, των της διδασκαλίας των διδαχών του Ιησού. Η περιγραφή του Νίμπουρ ε, είναι η εξής. Ένας θεός χωρίς οργή έφερε ε, ανθρώπους χωρίς αμαρτία σε ένα βασίλειο χωρίς κρίση μέσω ε, Μια ιεροσύνη ενό Χριστού χωρί ε, σταυρό. Όπω και στην ε, εποχή του Λουθύρου πριν από 500 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Χριστιανοσύνη χρειάστηκε να διαλέξει μεταξύ τη θεολόγια κρούση, δηλαδή τη θεολογία του Σταυρού, και τη θεολόγια, Γλώρια, δηλαδή τη θεολογία τη δόξα. Και τότε, στο ευρωπαϊκό σύστημα, πολλοί εκκλησιαστικοί ηγέτε συνεργάστηκαν με του τυράννου αντί ε, να πάρουν την πλευρά του της ε, θρησκείας. Ε, υπάρχουν ε, και στον ελεύθερο κόσμο όμως πειρασμοί. Πολλές πλούσιες εκκλησίες σε πλούσιες χώρες φαίνονται να ντρέπονται για το Χριστό και, οι παραδοσια... και τις παραδοσιακές βιβλικές χριστιανικές αξίες γενικότερα πολλοί κόσμος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια ότι, ώστε τα χριστιανικά σύμβολα να μην θίγουν ε, άλλες θρησκείες ή μη θρησκείες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παράδοξα ε, αποτελέσματα ε, να μην υπάρχουν πια σταυροί που να φοράει κανείς στο λαιμό του ή να μην υπάρχουν πια σταυροί στην εκκλησία σε διάφορες απεικονίσεις των εκκλησιών ή μερικές φορές δεν υπάρχουν καν σαν χριστουγεννιάτικα δέντρα στις ε, μεγάλες πλατείες των ε, μεγάλων πόλεων. Το έχουμε ακούσει αυτό. Ε, και δεν αναφέρομαι μόνο ε, στα χριστιανικά σύμβολα αλλά και στα Ιουδαϊκά και στα ε, μουσουλμανικά. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα πρόσωπο, μια πρόσωπη απεικόνηση της θρησκείας. Απομακρύνεται από το όραμα ε, του Αποστόλου Παύλου και δίνουν και πάλι χώρο στο μύθο. Επίσης υπάρχει κάτι ακόμη παγανιστικό είναι η αποκαλούμενη πολιτική χριστιανοσύνη όταν ε, η Εκκλησία υπηρετεί την πολιτική. Στην πολιτική χριστιανοσύνη ε, τα πολιτικά συμφέροντα συνδέονται με τα συμφέροντα της Εκκλησίας. Αν μια πολιτική ηγεσία αναλάβει ε, την εξουσία κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ένας, ε, μια πατεναλιστική προσέγγιση της πολιτικής Εκκλησίας. Μπορεί η Εκκλησία τότε να μην ε, αντιληφθεί καν πόσο στενούς δεσμούς έχει με την πολιτική εξουσία, ειδικότερα αν έχει υπάρξει καταστολή ή καταπίεση στο παρελθόν. Θα μπορούσα εγώ δηλαδή να σας δώσω και κάποια παραδείγματα από τη δική δική μου Η έλλειψη διαφάνειας και συνέχειας ε, στη χρηματοδότηση των εκκλησιών όπως επίσης και γενικότερα των οικονομικών της εκκλησίας ε, προσθέτει στην εξάρτηση των εκκλησιών ε, πολλές φορές ε, οι ηγέτες ε, αφήνουν στην πείνα τις ε, εκκλησίες και μερικές φορές θέλουν παρόλα αυτά να υπάρχει μια θρησκευτική λειτουργία που θα συνοδεύει κάποιες πολιτικές εκδηλώσεις και δεν είναι ωραίο για μια εκκλησία να έχει αυτόν τον άχαρο ρόλο. Ε, οι νεοφώτιστοι επίση έχουν και εκείνοι ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Μερικές φορές έχουν προσωπικές επιδιώξει και φιλοδοξίες. Ε, κάποτε στην Ουγγαρία, ε, κατά την κατάρρευση του σοσιαλισμού, ε, αναφερόταν κάτι που θα μπορούσε να επαναληφθεί για την περίπτωση αυτή, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόξιμο στο δρόμο για τη Δαμασκό. Δεν χρειάζεται να πει κανεί ότι αυτοί οι οπορτουνιστέ δεν είχαν ιδέα ότι αυτό που συνέβη στο δρόμο για την Δαμασκό δεν ήταν απόφαση του Παύλου, αλλά ήταν ε, ο ε, αναστηθής Χριστός και ότι ο Παύλος δεν ε, κατέληξε να είναι στην πλευρά των νικητών, αλλά των χαμένων. Στην, δεν, δεν ήταν στην λαμπερή πλευρά της υπόθεσης, αλλά στην σκιερή ήταν μάλλον η θεολογία του Σταυρού και όχι η θεολογία της δόξα. Η πολιτική χριστιανοσύνη έχει διάφορες μορφές. Στην Ανατολική Ευρώπη μπορεί να περιγραφεί για παράδειγμα μέσω ενός βιβλίου του Μάρτιν Σούλτσε Βέσελ ε, η εθνικοποίηση τη θρησκείας και ε, η ιεροποίηση του κράτους. In Eastern Europe την ε, Ανατολική Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ε, παραδείγματα από πολλές χώρες ε, στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, σας ανέφερα δύο διαφορετικά μοντέλα. Το ένα μοντέλο είναι κυρίαρχο στην Ανατολική Ευρώπη, το άλλο στην Δυτική όμως αυτή τη στιγμή ε, έχουμε την εμπειρία ενός, ε, μιας ανάμειξης των δύο και συμπερασματικά θα μπορούσα να πω να αφήσουμε τις εκκλησίες να είναι εκκλησίες, να αφήσουμε τις θρησκευτικές κοινότητες να είναι θρησκευτικές κοινότητες. να μην επιστρέψουμε σε ένα παγανιστικό κόσμο ε, με σύμβολο ε, την ε, βιαιότητα του Λευκού Ταύρου στην ελληνική μυθολογία και δεύτερον οι κυβερνήσεις ή άλλοι θεσμοί δεν θα έπρεπε να είναι πατερναλιστικοί με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικέ κοινότητες. Γι' αυτό όλοι όλοι μας ακούμε ε, τις κραυγές που μας λένε «Ελάτε να μας βοηθήσετε» είναι η, αυγή, είναι η κραυγή ε, της Ευρώπης ε, η οποία πρόκειται να ξεχάσει πώς να προσεύχεται, πώς ε, να... προς να τραγουδά και πώς να είναι των Κύριων. Μπορούμε να ακούσουμε αυτή την κραυγή. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις των ομιλητών δύο λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Μπορούμε να περάσουμε μέσω λοιπόν στη συζήτηση και θα ήθελα να ρωτήσω ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο για να θέσει κάποιο ερώτημα ή να κάνει κάποια παρέμβαση. Σας ευχαριστώ, θα κλείσω και τότε θα δώσω τις ευχαριστίες. Πρώτα θα ήθελα να σταθώ σε δύο συζητήματα που αναφέρθηκαν ε, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί εάν η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα, εάν παραμείνουμε ε, ως έχουν, αν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στο μέλλον. Και δεύτερον, είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε εν παρόλ, ε, θα είναι ο αντίκτυπο του Brexit. Πιστεύετε ότι το γεγονό ότι μια μεγάλη, ένα μεγάλο κράτος μέλος αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ε, θετικά ενθαρρύνοντας τα άλλα κράτη-μέλη ή ενθαρρύνοντας ακόμα τους πολίτες στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου να καταλάβουν καλύτερα ποια είναι η σημασία και τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. Σε ευχαριστώ. Επίσκοπος Αθανάσιος, εκπροσωπώ την Εκκλησία της Ελλάδος. Με χαρά άκουσα τους πολλούς φίλους ε, σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μεταφέρω ορισμένες ανησυχίες των Ελλήνων έχουμε προβλήματα. Επομένως, η προφανής απάντηση στο ερώτημά σας είναι η εξής. Εάν δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπης δεν θα χάσουν την εμπιστοσύνη που είχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό που υποτίθεται πως ε, συμβόλιζε και θα χαθεί αυτό το όραμα, αυτή η πεποίθηση ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια ευημερούσα και προοδευτική Ευρώπη. Η εν πάση περιπτώσει θα χαθεί σταδιακά. Δεύτερον, ακούστηκε ε, πολλές φορές η έκφραση μιας ανησυχίας για σημαντικές αξίες τις οποίες υποστηρίζουμε. Όμως, θα θέτω εγώ το εξή ερώτημα. Α κοιτάξουμε τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, ή τα τεράστια προβλήματα της που έχει δημιουργήσει η μεταναστευτική κρίση, οι οποίοι ε, αναγκάζονται να καταλήψουν τις αιστείες τους εξαιτία των κακουχιών που ε, ζουν σε αυτές, στις χώρες τους και αναγκάζονται να φύγουν. Ε, ρωτώ λοιπόν, ποιε είναι οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εφαρμόζονται σε όλα αυτά. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο έχω απευθύνει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανθρώπου που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, η απάντηση που λαμβάνω είναι ότι οι λύσει που δίνουμε είναι εμβαλωματικέ, γιατί στην πραγματικότητα οι ουσιαστικέ πολιτικέ δεν διαμορφώνονται τόσο στι Βρυξέλλε, όσο σε άλλα κέντρα λήψη αποφάσεων, η Ουάσιγκτον, τη Μόσχα και αλλού. Ε, είναι σημαντικό πάντω. Αυτό. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει την κατάθεση στη Μέση Ανατολή. Αυτό μου λένε, αυτό όμως εγώ δεν μπορώ να το μεταφέρω πιστικά στους δικούς μου συμπολίτες. Ίσως λοιπόν η Ευρώπη να προασπίζεται αρχές και αξίες οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τα συμφέροντα ή τις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον ή άλλων κέντρων λήψης αποφάσεων παγκοσμίω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξώσουμε το ανάστημά μας, γιατί να ακουστεί η φωνή της ε, Ευρώπης σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να δείξουμε στους πολίτες ότι δεν πρόκειται μόνο για λόγια, δεν έχει μόνο λόγια η Ευρώπη, η Ευρώπη αλλά επίσης ε, κάνει και έργα. Έχω άλλες τις παρεμβάσεις. Παρακαλώ, εστέ ε, σύντομη. Έχει επίσκοπε Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, που υπόθηκαν, η προσφυγική κρίση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στην Ελλάδα αφορούν την αξιοπιστία της Ευρώπης. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτές τις κρίσεις, δεν είμαστε πλέον αξιόπιστοι. Τώρα για τα δύο ερωτήματα. Το θέμα της αλλαγής. Ναι, πρέπει να αλλάξουμε, είναι η απάντησή μου. Πρέπει να αλλάξουμε επίσης γιατί αλλάζει και ο κόσμος. Ακούσαμε να αναφέρεται η ψηφιοποίηση, η ατομικότητα, όταν έχουμε μεγάλη αλλαγή του πολιτισμού και δεν γνωρίζουμε επακριβώς πώς αλλάζει ο πολιτισμός και πώς η πολιτισμική αλλαγή επηρεάζει την πολιτική, τη δημοκρατία κλπ. Ε, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της αλλαγής. Να την έχουμε υπόψη μας. Και να παλέψουμε για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Το Brexit τώρα. Δεν ξέρω τι μορφή θα έχει. Βλέπετε παίζουν ρόλο διάφορες δυνάμεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Κάποιοι θέλουν ακόμα στενότερη ένωση και άλλοι λένε φτάνει, ως εδώ. Πιστεύω το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα κινηθεί. Αν πραγματικά δει τα πραγματικά προβλήματα των απλών ανθρώπων και βρει απαντήσεις. Τότε έχουμε πραγματικά πιθανότητες. Πραγματική πιθανότητα. Ευχαριστώ. Εδεσιμότατε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις στα δυνατά αυτά ερωτήματα της Αντιπροέδρου της κ. Μακίνες. Ελπίζω να μην κάνετε, να μην κάνετε το τίποτα, να κάνετε κάτι δηλαδή. Είμαι ιστορικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε λόγω ανάγκης συμφιλιώσεως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν δείτε πόσο περίπλοκα ήταν τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα κομμάτι του προβλήματος ήταν η αδράνεια. Να μην γίνεται κάτι. Άρα αυτό δεν είναι λύση το να μην κάνουμε κάτι. Το Brexit τώρα θα αποβεί κάτι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η μορφή του Brexit. Και από ό,τι βλέπω, ακόμα κανείς στις Βρυξέλλες ή στο Westminster δεν γνωρίζουν ακόμα. Ε, συνεχίζεται η συζήτηση. Υποτεθεί το ότι θα είναι ένα καλό Brexit όπως το αποκαλούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Good Brexit. Που θα είναι καλό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τότε ίσως αυτό να παίζει ρόλο και για την ευρύτερη Ευρώπη που ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος ο Σεβασμιότητος Άλτριτς. Η Ενωμένη Ευρώπη δίνει πολλές επιλογές που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο τι μορφή θα έχει ευρύτερη Ευρώπη. Δεν πίστευα να το πω αυτό. Ίσως ένα καλό Brexit, ίσως να συμβάλλει σε αυτή την ευρύτερη Ευρώπη. Ένα καλό Brexit. Ιαν Άλμπρεχτ, το συνάδελφο. Από την Πολωνία, είμαι ευρωβουλευτή, Δύο ερωτήσει. σχόλιο και ερώτηση. Σχόλιο πρώτα. Μιλώντα για διεύρυνση. Δεν αφορούσε χρήματα διεύρυνση για τη χώρα μου. Ήθελε η χώρα μου να ανήκει στο δυτικό πολιτισμό. Μετά άλλαξε η κατάσταση. Βασικός λόγος ήταν να ενταχθούμε στην ευρωπαϊκή νοοτροπία και την κουλτούρα. Εγώ είμαι καθολικός. Ζω σε ένα μέρος της Πολωνίας που επηρεάζεται πολύ από τη Λουθυρανική Εκκλησία πήγα ε, στον ετασμό της 500ης επαιτίου της μεταρρύθμισης και στην προσευχή είπα να προσευχηθούμε για τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες. Είναι πολύ σημαντικό να μην συγκεντρωθούμε μόνο επί των προσφύγων, αλλά να προσευχόμεθα για όλους που έχουν την ανάγκη μας. Και οι οικονομικοί μετανάστες είναι άνθρωποι με ανάγκες. Να πω κάτι είναι ήδη προκλήσεως. Και κάτι που είναι δύσκολο. Το προκλητικό. Αν αυτό το πάνελ είναι υπέρ ενδεχόμενης αλλαγής της συνθήκης. Φαντάζεστε τη συζήτηση για την νέα αλλαγή, η μετατροπή της συνθήκης. Θυμόστε τη συζήτηση για την ε, θέμα της δημοκρατίας, Democracy Day. Αν ξαναρχίσει η διαπραγμάτευση συνθήκη, αυτή του είδους η συζήτηση θα αλλάξει. Έχουμε διαφορετικό κόσμο σήμερα. Αν αλλάξει συνθήκη, χρειαζόμαστε κάποια σχετικά στοιχεία με αυτό που συζητούμε. Δεύτερον, εμείς που συμμετέχουμε στο διαθρησκευτικό διάλογο αντιμετωπίζουμε προβλήματα καθορίζοντας ποια είναι η θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη, η ανεξιθρησκεία. Τι έχετε να προτείνετε σε εμάς τους πολιτικούς Πώς να αντιληφθούμε την ανεξιθρησκεία, την ελευθερία της σχετικής έκταση σήμερα. Ορίστε, κυρία μου, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο εκ νέου. Στο ερώτημά σας, τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρία σημεία δεν αναφέρθηκαν. Περισσότερη ειλικρίνεια χρειάζεται σίγουρα από πολιτικού. Γιατί μπορεί να κάνει η Ευρώπη και τι δεν μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Κατά παρελθόν νομίζω δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις που δεν ετηρήθησαν και απογοήτευσαν πολύ τους πολίτες. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στο μέλλον. Μετά, να πλησιάσει η Ευρώπη τους πολίτες και να διδοθεί αισιοδοξία για το μέλλον. Αυτά τα δύο στοιχεία, οι εκκλησίες και οι θρησκευτικέ οργανώσεις μπορούν να παίξουν ρόλο. Διότι είμαστε κοντά στα μέλη μας και μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον. Και να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ του πολιτικού κόσμου και του λαού. Και κάτι άλλο που δεν τονίστηκε και δεν συζητήθηκε επαρκώς. Το μεγάλο θέμα. Πώς θα αντιμετωπίσουν τους όσφυγες που αναφέρεται και τους οικονομικούς μετανάστες. Τώρα που τονίζεται το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που έχει αποτελματωθεί στο Συμβούλιο. Εμείς σαν εκκλησίες σε οικουμενικό πλαίσιο μπορούμε να παίξουμε δραστήριο ενεργό ρόλο για να ξεπεραστούν στερεότυπα και παρεξηγήσεις για τους αλλοδαπούς και να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό και για την αξιοπιστία της Ευρώπης και για το μέλλον της. Πρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα εκεί, δημιουργώντας νόμιμες ε, διαδρομές για τους ε, πρόσφυγες. Να μην καταδικάζονται σε πνιγμό στη Μεσόγειο αυτοί οι πρόσφυγες. Χρειάζεται επιμερισμός των ευθυνών. Να συμμετέχουν εξανατολών και εκδισμών. Και θέλουμε ως εκκλησιαστικοί φορείς και εκκλησίες να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ορίστε. Πόσοι θέλουμε να μιλήσουν, να πάρουν το λόγο. Έχουμε δύο που θέλουν να πάρουν το λόγο εκεί. Α, και εσείς. Τρεις. Ισαμπέλ Μαφάρ του κινήματος Φοκολάρη. Τι κάνουμε. Μιλήσαμε για την παιδεία, πρωτοβουλίες των πολιτών, εμπειρία θρησκευτικών κοινοτήτων που παρίστανται εδώ, στο διάλογο, πέρα από το θέμα της ποικιλομορφία. Μιλήσαμε και για το πρόγραμμα Έρασμος που συνέβαλε ούτω ώστε οι νέοι οι Ευρωπαίοι, νέοι Ευρωπαίοι να έχουν ένα φυσικό ορίζοντα της Ευρώπης και όχι εθνικό ορίζοντα. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε και ενθαρρύνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν στους νέους της Ευρώπης που πολύ συχνά μεγαλώνουν σε ένα πλαίσιο που έχουν ψευδή εικόνα είτε κοσμικότητας είτε ουδετερότητας να εκμεταλλευτούν ε, την εμπειρία και τη σοφία που εκφράστηκε εδώ στη συζήτηση και να έχουν σαν φυσικό ορίζοντα μια Ευρώπη στην οποία η ποικιλομορφία της πίστης και των θρησκειών είναι κάτι επικοδομητικό και να θεωρηθεί σαν θέμα συνεργασίας ενεργού ε, για την ειρήνη και όχι απλώς μια ανοχή ή που είναι η ιδιαιτερότητα οδηγεί σε πρόθεση της ειρήνης περισσότερο από τη θρησκεία. Θα πρέπει και μη θρησκευτικοί φορείς συμμετάσχουν σε αυτό. Αλλά σε τεράστιο επίπεδο, όπως και έγινε για το Έρασμος, πάρα πολλοί νέοι, να υπάρχει σε τεράστια κλίμακα ένα πρόγραμμα, να μπορούν να συμμετέχουν και οι νέοι. Είναι πάρα πολύ θεμελιώδε αυτό το θέμα της παιδεία. Ευχαριστώ. Μίκολα, πρόεδρος του μέλλοντο για την Ευρώπη οι πολιτικοί συζητούν, προτείνουν μέσα πολιτικές λύσεις ή οικονομικές λύσεις. Οι εκπρόσωποι ε, των θρησκειών ε, και των ε, ηθών μιλούν για αξίες, μιλούν για ιερές αξίες, του πώς εφαρμόζονται. Πρέπει οι πολιτικοί και αναφέρομαι στην ε, παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Χόλεριχ. Η κρίση της Ευρώπης είναι κρίση αξιοπιστίας και μια κρίση αξιοπιστίας ε, αφορά όλες τις αρχές και για να βγει κανείς ε, από την κρίση αυτή πρέπει οι αρχές, όλες οι αρχές να καταστούν αξιόπιστες και για να καταστούν αξιόπιστες πρέπει να είναι συνεκτικές, να παρουσιάζουν συνοχή. Δεν έχει νόημα να ε, διακηρύττει κανείς ε, όταν τελικά ε, εσωτερικά δεν εφαρμόζει τις αξίες που προτείνει στους έξω να εφαρμόσουν. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν στις, τις αξίες να τις δούμε λίγο καλύτερα και να προσπαθούμε καταρχάς να τις εφαρμόζουμε εντός των πολιτικών θεσμών και επίσης οι ε, θρησκευτικές αρχές ε, θα έπρεπε να ασχολούνται λίγο περισσότερο την πτυχή της οργάνωσης της κοινωνίας. Ποιες είναι οι λύσεις δηλαδή που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να βελτιωθούμε. Για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματα στο φάκελο που λάβατε όλοι έκανε μία προσπάθεια και προτείνουμε για παράδειγμα να ε, γίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πραγματική κυβέρνηση που θα εκλέγεται και που θα είναι υπεύθυνη και ε, υπόλογος. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε και οι εκπρόσωποι των θρησκειών να κάνουν και εκείνοι να συνεργαστούν στενά και αποτελεσματικά ε, να συμμετέχουν σε αυτήν τη συζήτηση που δεν μπορεί να είναι μια συζήτηση μόνο μεταξύ πολιτικών. Πρέπει το ηθικό κομμάτι, για να το πω, να το πω έτσι, ε, της Υπήρου μας ε, να πάρει στα χέρια του ε, ε, το πρόβλημα. Η αξιοπιστία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα ζήτημα συνοχής. Αν δεν είμαστε συνεκτικοί με αυτό που εμείς προτείνουμε προς τα έξω, στους άλλους, αν εμείς δεν ακολουθούμε τους ίδιους μας τους κανόνες, υπάρχει ο κίνδυνος να, συνεχίσουμε να μιλάμε ε, χωρίς ουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ εμπνευστική αυτή η συζήτηση. Τελευταία παρέμβαση. Ρισελ Μπαϊάννη από ε, την... Ε, από το Behind National Community. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο καθένας επισημαίνει μία πτυχή του μέλλοντος της Ευρώπης και εγώ θα ήθελα να πω προσπαθώντας ε, να συνοψίσω κάπως και να δω ε, τι υπόθηκε πάνω κάτω σε όλες τις ε, παρεμβάσεις είναι ότι η μοίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή του υπόλοιπου κόσμου. το πλεονέκτημα του ενός ε, επιτυγχάνεται καλύτερα από το πλεονέκτημα όλων. Είναι δύσκολο λοιπόν ε, να ε, ασχολούμαστε με το πλεονέκτημα του ενός χωρίς να ασχολούμαστε με το πλεονέκτημα του άλλου γιατί το πλεονέκτημά μας θα είναι πολύ περιορισμένο. Οπότε να δούμε πρώτα τα του οίκου μας και να βάλουμε τάξη στο δικό μας το σπίτι, να δούμε ότι η λογική αυτή δεν ισχύει διαφορετικά. Ε, όσο δύσκολο και ξεζητημένο και αν ακούγεται αυτό, σημαίνει ότι οι πολιτικές μας, ε, και το βλέπουμε όλο και περισσότερο, οι οικονομικές πολιτικές, ε, πολιτικές μετανάστευσης, όταν ε, σκοπό έχουν μόνο να δημιουργήσουν ευημερία σε ένα μόνο μέρος του κόσμου, δεν μπορούν να δημιουργήσουν ευημερία στο υπόλοιπο, ε, στον υπόλοιπο κόσμο, δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν την ευημερία ούτε στο δικό τους κομμάτι του κόσμου. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχω μερικά λεπτά στη διάθεσή μου για να προσπαθήσω να συνοψίσω κάπως αυτό που, αυτά που μόλις ακούσαμε νομίζω ότι Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε πολύ με οικονομικά ζητήματα. Πρέπει να πει κανείς ότι ε, υπήρξε μια κρίση που ήταν πάρα πολύ σκληρή, πολύ δύσκολη, δυσκολότερη για κάποια τμήματα της Ευρώπης όχι όμως υποχρεωτικά αυτοί που ήταν η περισσότερο ορατοί, γιατί η κρίση στο εσωτερικό κάθε χώρας ε, έπληξε ε, πολύ κόσμο, ακόμη και αν δεν έγινε απολύτω αισθητό αυτό. Όλη αυτή η αρνητική στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει και από εκεί, από τη μη κατανόηση του γεγονότος ότι το γεγονό του να είμαστε μαζί ε, είναι, έχει σκοπό να αποφύγει τα χειρότερα. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για μερικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Όλες ε, οι χώρες παρόλα αυτά συνεισέφεραν στο να αποφευχθεί το χειρότερο για την ε, Ελλάδα, ε, δραματικές εξελίξεις, ακόμη και ως προς τους πρόσφυγες. Εμείς καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά προσπαθούμε να συνεργαστούμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε από κοινού και σε πολλές περιπτώσεις ε, υπήρξαν αποτελέσματα στη χώρα μου για παράδειγμα, στην Ιταλία δεν βλέπουμε για την ώρα την μείωση των αφήξεων στην Ελλάδα όμως υπήρξε μείωση των αφήξεων χάρη σε μέρη και στην κοινή προσπάθεια νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι πολύ σημαντικός είδαμε ότι στη Γαλλία ήταν επαρκές να αλλάξουμε το λόγο ε, την, ε, για την Ευρώπη για να υπάρξει και πάλι μια νέα, καλύτερη, θετικότερη στάση των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι για όλους, γιατί είναι πολιτικό ζήτημα, είναι κάποιοι που είναι υπέρ και κάποιοι που είναι κατά. Αν όμως όλοι οι πολιτικοί, στο πλαίσιο του δικού τους ρόλου, οι εκπρόσωποι των ε, πολιτών ε, στο δικό τους ρόλο, ε, των θρησκευτικών κοινοτήτων επίσης, μιλούν θετικά, έχουν ένα θετικό λόγο όχι να επενέσουν υποχρεωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξουν πόσο σημαντικό είναι να συνεργαστούμε για το μέλλον της Ευρώπης, υπάρξουν πράγματα που θα είναι θετικά και δεν θα χρειαστεί να τα αλλάξουμε και πράγματα που θα χρειαστεί να αλλάξουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε ε, από κοινού και μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Αν αν δεν θέλουμε να βγούμε από την ιστορία του μέλλοντος, πρέπει να παραμείνουμε από κοινού, ε, ε, να συνεργαστούμε, όπως είπε ένας φιλόσοφος. Και νομίζω ότι εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε ε, και θέλουμε να μάθουμε και πολλά σε άλλους, ε, στον υπόλοιπο κόσμο έχουμε μια ιστορία θρησκευτικών πολέμων αρκετά σημαντική. Ακούγοντας λοιπόν εσάς και ακούγοντας ο ένας τον άλλον κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα μια θρησκευτική ανεκτικότητα η οποία είναι ε, άνευ προηγουμένου στον κόσμο. Βέβαια δεν μπορεί να επαγρυπνά ποτέ κανείς, δεν είναι όλα ε, και εκτιμένα ε, Δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε καν αυτό είναι και εκτιμένο Είναι όμως μία αξία και ένα παράδειγμα για άλλα τμήματα της Ευρώπης, όπου ακόμα σήμερα ε, υπάρχουν πόλεμοι για θρησκευτικούς λόγους. Ο πόλεμος στον Ισλαμικό κόσμο και εναντίον της Ευρώπης βεβαίως, όπως έγινε μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών ε, ε, αυτό έγινε πρώτα σε εμά και μετά στο Ισλάμ. Ε, το, το θέμα αυτό λοιπόν της ανοχής που δείχνουμε εμείς σε όλες τις θρησκείες είναι κάτι που μπορεί να, από αυτό να μάθει ο υπόλοιπο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευρυνθεί γιατί το μέλλον μας θα είναι πολύ θρησκευτικό θα υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, θρησκείες ε, και ομολογίες. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όταν όμως έχουμε αξίες στους θεσμούς μας, στις συνθήκες μας, στον πολιτισμό μας και τις έχουμε αυτές τις αξίες της θρησκευτική ανοχής, ε, τότε μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές. Και νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη του δική σας βοήθειας για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ε, ε, ότι το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι ένα σύνολο αξιών πολύ σημαντικών ε, για τη ζωή μας και για το μέλλον μας. Μόνο από κοινού μπορούμε να υπερασπιστούμε τις αξίες αυτές, να τις εφαρμόσουμε, να τις κάνουμε να έχουν αξία και παράλληλα να είναι και μία ισχύς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υπάρξουμε ε, στον μελλοντικό κόσμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό το διάλογο, τη συζήτηση και νομίζω ότι αν πρόκειται να ξαναρχίσει συζήτηση για τις συνθήκες θα το κάνουμε. Αργά ή γρήγορα. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις αξίες, ε, στις συνθήκες το είχαμε αφήσει αυτό κατά μέρο ε, από το φόβο ε, ότι δεν θα ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι. Όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να το λάβουμε πολύ σοβαρότερα υπόψη, να ε, δώσουμε στου Ευρωπαίους ένα όραμα, όπως όλοι είπατε, ένα όραμα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορούμε να το κάνουμε αν σε αυτή τη συζήτηση για την αναθεώρηση των συνθήκων συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών, της οποίας μεγάλο κομμάτι είστε κι εσείς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Δεν θα κάτσουμε μεταξύ μας ε, ε, και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα, να τα αποφασίσουμε και να καταλήξουμε. Πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες. Εντάξει, προφανώς επισήμως ε, θα πρέπει να ε, κάνουμε τις αλλαγές όπως πρέπει για να σεβαστούμε τους κανόνες των συνθήκων. Σας αφήνω λοιπόν να προβληματιστείτε, να το σκεφτείτε περαιτέρω, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μάθαμε από την κρίση ε, και από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε και σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λοιπόν το μέλλον, να το ατενίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρέσο. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιε μικρέ ε, καταληκτικές παρατηρήσεις, αλλά πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω αν ήθελε κάποιο από του ομιλητέ του πάνελ το λόγο. Βεβαίω. ελάτε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ουγγρικά. Σπάνια έχω τη δυνατότητα σε διεθνή συνάντηση να μιλώ ουγγρικά, επομένως θα το ξεπίσω. Με χαρά άκουσα, με πολύ ενδιαφέρον και χαρά άκουσα τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις της κυρίας Μπερεσό. γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις πράγματι στην ε, Ουγγαρία. Ε, όταν εγώ ε, προετοίμαζα το ταξίδι μου, υπήρξαν άνθρωποι στην Ουγγαρία που μου είπαν «Α, τώρα στις Φρυξέλλες που θα πας εκεί είναι μακριά, δεν έχει χαθεί η χριστιανοσύνη από αυτή την πόλη» κτλ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν σε αυτούς, τους, αυτόν το, τη συζήτηση, σε αυτόν τον διάλογο. Ε, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της μεσαιωνικής σκέψης που θεωρεί ότι η Εκκλησία ή η θρησκεία θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά από την άλλη εμείς στις ανατολικές χώρες έχουμε και την εμπειρία του περίοδου του κομμουνισμού που κατάφεραν οι εκκλησίες μας να επιβιώσουν και έχουμε πολύ έντονα ακόμα τις αναμνήσεις από εκείνη την εποχή που η ύπαρξη ακόμα και των θρησκειών ήταν κάτι το απαγορευμένο να αναφερθεί. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε αυτά τα δύο άκρα. Οι εκκλησίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης βασιζόμενες στην αρχή του ανθρωπισμού που τις διέπει όλες πολύ συχνά οι εκκλησίες στις χώρες μας ε, αναπτύσσουν συνεργασίες με μη κυβερνητικές οργανώσεις και, και, και υποστηρίζουν κινήματα αλληλεγγύης ή βοήθειας ή αρρωγής. Υπάρχουν λοιπόν πολλών διαφορετικών λογιών οργανώσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. η βοηθειας η αρρωγης υπαρχουν λοιπον πολλων διαφορετικων λογιων οργανωσεις οι οποιες μπορουν να βοηθησουν στην αντιπετώπιση των κοινωνικων προβληματων η καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, της κοινωνίας είναι σημαντικότατος ε, ρόλος που ε, αναλογεί σε κάθε εκκλησία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι δυνατόν να, δεν είναι προσβάσιμα για τις θρησκευτικές κοινότητες ή για τις εκκλησίες. Λαμβάνοντας υπόψη του σημαντικό ρόλο που έχουν οι εκκλησίες να παίξουν, να διαδραματίσουν, ίσως θα είχε μια αξία να σκεφτούμε το ενδεχόμενο ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια να μπορούν να διαθέσιμα και σε αυτές. Τα τελευταία δέκα χρόνια εγώ προσπαθούσα, ε, ήμουν ουσιαστικά νομαδικός. Ε, γνώριζα πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Στο χώρο των αραβικό, τον ισλαμικό, στη Συρία ιδιαίτερα, ξεκίνησαν πολίτες να πιστεύουν στις ευρωπαϊκές αρχές. Βεβαίως δεν τις αντιμετωπίζουν, δεν τις βλέπουν ως κάτι γεωγραφικά εντοπισμένο. Ε, τις ενστερνίζονται ως αρχές. Στις επισκέψεις που έκανα στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια διαπιστώνω μια διαφορετική δυναμική. Υπάρχει μια αίσθηση των πολιτών ότι απειλούνται γεωγραφικά και τώρα προσπαθούν να, χρησιμοποιήσουν τις αξίες τους ως όπλο για να υπερασπιστούν τη γεωγραφική τους επικράτεια θέση. Πρέπει κατά την άποψή μου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυναμική στην Ευρώπη. Υιοθετώντα μια προσέγγιση η οποία δεν, δεν, δεν, δεν ορίζει τις ευρωπαϊκές αξίες με βάση τη γεωγραφική τους, τον γεωγραφικό του εντομισμό, γιατί δεν έχει νόημα ε, κατά τη δική μου άποψη. Και εγώ είμαι, αισθάνομαι Ευρωπαίος και ταυτόχρονα μουσουλμάνος. Το ηθικό μου χρέος είναι να συνεργάζομαι έτσι ώστε να αναλάβουμε δράση από κοινού για να προασπίσουμε αυτές τις αξίες που μας επιτρέπουν να συνεπάρχουμε. ως το, προς, την ταυτότητα ε, δεν καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε ούτε μεταξύ μας οι μουσουλμάνοι, ούτε εγώ με τους μουσουλμάνους αδελφούς μου. Ε, σε, άλλες, λοιπόν, σε άλλους πολιτισμούς το ζήτημα της ταυτότητας τίθεται διαφορετικά. Σε ορισμένες γλώσσες δεν υπάρχει καν ο, ο, τρόπος να, να, να, θέσει το ερώτημα με την, με, το, με την ε, διατύπωση ποιος είμαι. Θα έλεγε κανείς τι, τι κάνω, τι πράττω. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια φιλοσοφική συζήτηση, την οποία ίσως καλύτερα να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Να το σκεφτούμε. Καλό θέμα. Τελευταία λέξη τώρα, τελευταία σας παρέμβαση, Μπορείτε να μιλήσετε και στη γλώσσα σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας μιλήσω γοδελικά και λυπούμε. Προσπαθώ να μάθω γαλλικά. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε, εκ μέρους όλων μας. Εκ μέρους της ε, κοινωνίας των τελευταίων θρησκειών που εκπροσωπούνται, τολμώ να πω, είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος. Έχω παραστεί σε διάφορους διαλόγους διαφόρων ειδών. Έχω έρθει στις Βρυξέλλες για αυτούς τα τελευταία χρόνια. Αυτός ήταν ο χρησιμότερος. Αυτό να το εισακούσετε, αυτού του είδους η πρακτική ανταλλαγή απόψεων είναι απελπιστικά, τεραστίως σημαντική αν μπορώ να το πούμε αυτό. Και ε, το αφορά τις σκεφτικές κοινότητες διότι ε, αγαπάμε το Θεό και ο Θεός μας φροντίζει. Κοιτάξτε, ειλικρινά αυτό είναι το συμπέρασμα, η κατάληξη. Ίσως διαβάσατε την <laughs> παρέμβασή μου. Ε, ίσως επειδή είμαστε και γραφικά γείτονες με καλύψατε. Είχα κάποιες σκέψεις, αλλά νομίζω ότι αυτό το σχόλιο το καταληπτικό ήταν ισχυρότατο. Εν συντομία, τρία πράγματα μου έρχονται από τη συζήτηση. Η Ευρώπη δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται ε, τροφοδότηση, αλλαγή και θέλετε να συμμετάσχετε στην αλλαγή και θέλουμε και εσείς να είστε ένα κομμάτι αυτής αλλαγής. Δεύτερον, ο Αρχιραβίνος αναφέρθηκε στην ισορροπία ευθυνών και δικαιωμάτων. Καμιά φορά όταν μιλώ σε πολίτες είμαι άμεσα εκλεγμένη εκπρόσωπος, άρα αφιερώνω τη ζωή μου στους εκλογείς μου. Καμιά φορά όταν με αφισβητούν και μου λένε τι δεν κάνει η Ευρώπη είσαστε όλοι μέλη της ελίτ και γραφειοκράτες, πρέπει να τους ε, προκαλέσω απατώντας και να πω με κάθε σεβασμό εγώ έχω τεράστιες ευθύνες εδώ. Προσπαθώ να ηγηθώ. Εσείς σαν πολίτες έχετε τεράστιες ευθύνες να ανήκετε στην προσπάθεια οικοδομήσεως ε, ενός εγχειρήματο ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους λόγους που αναφέρατε όλοι. Ποτέ δεν λιώνει η δουλειά μας, είναι το τρίτο σχόλιο μου. Και γι' αυτό σίγουρα αυτό είναι ένα κομμάτι ενό διαλόγου που θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσει η επαφή μαζί σα και ελπίζουμε και εσεί να κοβεντιάσετε μαζί μα. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίω του Προέδρου, που ήταν πολύτιμοι στο να καθοδηγήσουν τη συζήτηση και για τα παρόντα μέλη. Η παρουσία σα είναι ιδιαίτερα σημαντική και άκρο ευπρόσδεκτη και για μένα, αλλά και για εκείνου που ήρθαν να μα μιλήσουν. Και βεβαίω, μετά από κάθε διάσκεψη και ενδελεχή ε, συζήτηση πρέπει να υπάρξει μια δεξίωση όπου και εκεί μπορούμε να κουβεντιάσουμε μεταξύ μα πιο ανεπίσημα. καλό όλους τους προσκεκλημένου να πάμε κάτω έναν όροφο, χρησιμοποιείτε τη σκάλα ή του ανελκυστήρες, σα βοηθήσω συνάδελφοι να σα πω ότι έχουμε κόσερ και χαλάλ τρόφιμα, φαγητά, στον πέμπτο όροφο του κτηρίου αυτού και θα σας βοηθήσουν, θα σας καθοδηγήσουν πώς να πάτε εκεί. Κλείνοντας, είναι η πρώτη μεγάλη μου συζήτηση σε επίσημο πλαίσιο μαζί σας. Είπα από την αρχή ότι με προσήλκησε πολύ ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην αίθουσα και παρέμεινε στην αίθουσα, αυξήθηκε αυτό το κλίμα, το ευχάριστο συζήτηση. Όλοι παλεύουμε να κάνουμε το σωστό μέσω τη συζήτηση. Αλλά μα βοηθάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, προσβλέπω στην δεξίωση. Ευχαριστώ όλου. Καλό σα βράδυ.